Okay, if uh, people could settle down, um. Καθίστε, παρακαλώ. Τα τυπικά πρώτα. Πρώτα απ' όλα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Καλώς. Συνέχεια έγκριση των πρακτικών. Έχουμε πρακτικά το συνεδριάσεων 28 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου, το 10-13 Φεβρουαρίου, 13 Φεβρουαρίου πάλι και 17 Φεβρουαρίου του 2014, έτσι. Εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Καλώς. Ανακοινώσεις και ενημέρωσή σας για τους ε, τριμερείς διαλόγους. 25 Φεβρουαρίου είχαμε τον τελευταίο τριμερή διάλογο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και έχουμε και τις διαπραγματευτικές έντολες και μια επιβράδυση των διαπραγματεύσεων. Ήταν βέβαια μεγάλη απογοήτευση για μας, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι είχαμε, μια, είχαμε δώσει μια ελαστική εντολή, αλλά φαίνεται ότι εξαφανίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Η γενική προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το Ταμείο Νιέου Μηχανισμού Καθάρισης. Επίσης, συζητήθηκε η συνεισφορά, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου αυτού και ο επόμενος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στις 4 Μαρτίου. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για τις πληρωμές, τρίτης τριμερής διάλογος έγινε στις 26 Μαρτίου. Επιτέχθη κάποια πρόοδο στον τομέα των κυρώσεων και των αρμοδίων αρχών και μπορεί να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός όσον αφορά τη διαφάνεια, την πρόσβαση και το διασυνοριακό switching. Υπάρχουν άλλοι δύο τριμερείς διάλογοι 13 και 20 Μαρτίου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο να πετύχουμε συμβιβασμό κατά τη διάρκεια αυτής ακόμα της εντολής. Ε, τώρα, αποζημιώσει. Δεύτερο τριμερή διάλογο έγινε στο Στρασβούργο. Εκεί προχωρήσαμε σε διάφορα σημεία. Μεταξύ άλλο, τα επιπλέον τέλη, άρθρα 12 με 15, διάδραση ανάμεσα στα πρόστιμα και το μέγεθος της ζημιάς και υπάρχουν και κάποιες γενικότερες ιδέες για συμφωνία όσον αφορά την κοινή ευθύνη που είναι το άρθρο 11. Συμφωνία πάντως μπορούσε να βρεθεί και για το closure evidence που είναι το άρθρο 6. Εξαρτάται βέβαια κάπως από τις εθνικές συμφωνίες και το άρθρο 9. Περιμένουμε να δούμε πότε θα μπορούμε να έχουμε μέσα Μαρτίου μάλλον έναν επόμενο τριμερή διάλογο για να πετύχουμε και συμφωνία πάλι για την θητεία αυτή. 5. Μετά τις συνομιλίες που είχαμε τα τρία θεσμικά όργανα, υπάρχει κάποια συμφωνία για γραπτή διαδικασία. 26 Φεβρουαρίου δεν χρειάστηκε ε, συμβούλιο εκεί. Πρόκειται για τις καταχρήσεις στην αγορά και για τις κυρώσεις Συμφωνία επί των αμοιβών επίσης. Και είδαμε τι, ποιοι καλύπτονται από την ρύθμιση αυτή για τις αμοιβέ usage όταν κάποιες αρμοδιότητες δίνονται σε τρίτα μέρη. Βάσει του άρθρου 17 θα γνωμοδοτήσουμε με τον ε, συνήθι τρόπο όταν θα έχουμε τελική επιβεβαίωσε από το Κορεπέρο ότι έχουν συμφωνήσει με το κείμενο. Στην ε, σύνοδο του Απριλίου θα τεθεί αυτό. Στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Τι άλλο, Κέι, έχεις πρόβλημα. Α, να Τώρα έχουμε νέα διαβούλευση όσον αφορά τον Εμμύρ. Βάσει το άρθρο 17 όσον αφορά τον διάλογο όπου καταλήξαμε στις 14 Ιανουαρίου με συγγετή τον Μάκος Φέβερ. Το Συμβούλιο μας επιβεβαίωσε στις 19 Φεβρουαρίου ότι εγκρίνεται η θέση του Κοινοβουλίου εφόσον το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με το συγκεκριμένο κείμενο. Ο εισηγητής, αν θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Τώρα, Μάρκος, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ακόμα και αν η υπόθεση αυτή η αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της ρυθμίσης αυτή για τις αγορές. Δύο χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα μπορούσε και νωρίτερα μάλιστα, αλλά το Συμβούλιο καθυστέρησε. Είχαμε λοιπόν διαπραγματεύσεις, τριμερείς διαλόγους, έξι μήνες. Τεράστια βέβαια πρόκληση ήταν αυτή που είχαμε μπροστά μας, γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω όλη τη διαπραγματευτική ομάδα και όλους τους συνεργάτες για την πολύτιμη βοήθειά του και τη γραμματεία της Επιτροπής και τις πολιτικές ομάδες. Χάρη σε καταφέραμε να έχουμε κοινό μέτωπο στις διαπραγματεύσεις αυτές και μπορούμε να είμαστε περήφανοι που 90% περίπου των συμφωνιών με το Συμβούλιο είναι ακριβώς αυτό που ήθελε και το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Συνεπώς η επιτυχία είναι μεγάλη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και σας ζητάω να εγκρίνετε το αποτέλεσμα αυτό και να το υποβάλλετε προς ψήφιση στην Ολομέλεια ως έχει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος το άρθρου 17. Μύθιτ και μύθιτ προς ψηφοφορία. τάσω στις χειρός, ότι συμφωνείτε να πάει στην Ολομέλεια δηλαδή. Είναι κανείς κατά, αποχές, καλώς. Ωραία. Θα υποβληθούν στην Ολομέλεια τα κείμενα αυτά και στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου θα ψηφίσουμε. Μετά βέβαια κάποιες μικρές γλωσσικές διορθώσεις στο κείμενο που βέβαια μπορεί να ανοίξει, μάλλον όχι, όχι, τίποτα δεν θα ανοίξει, έτσι θα πάει. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελάχιστε αυτές οι διορθώσεις. Τώρα, την ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε και όσον αφορά το CFDR. Υπήρξε συμφωνία τριημερού διαλόγου στις 18 Δεκεμβρίου, Ο υπόθηκε ότι στις 9 Ιανουαρίου και 26 Φεβρουαρίου θα προχωρούσαμε εν ώψη της επιστολής Κορεπέρ. Και για πες μας. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες. Ήταν πολύ τεχνικό το θέμα και οι τριμερείς διάλογοι. Όλοι λοιπόν όσοι βοήθησαν, οι σύμβουλοι λοιπά, Τους είμαι ευγνώμων για το χρόνο που διέθεσαν προκειμένου να καταφέρουμε να καταλάβουμε τι συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο. Δεν ήταν εύκολο, σας διαβεβαιώ. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Μας δίνει πάντως ε, κάτι πολύ γερό στα πλαίσια της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Εντοπίστηκαν βέβαια κάποιες ασυμβατότητες που νομίζω όμως ότι στο μεταξύ διορθώθηκαν. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί απρόσκοπτα να προχωρήσει σε αυτά τα οποία ζητάμε με την νομοθεσία. Και ελπίζω όλοι να υπερψηφίσουν. Ευχαριστούμε πάλι Βάση το άρθρο 17 διανατάσσεως τη χειρός, αν συμφωνείτε με το κείμενο να προθεθεί στην Ολομέλεια. Κατά. Αποχές. Ωραία. Πάλι στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου θα έχουμε αυτό το θέμα. Μάριο τώρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έπρεπε έτσι καλώς να ξεκινήσουμε κανονικά τις εργασίες μας. Είμαστε στον τελευταίο νομισματικό διάλογο για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Σήμερα λοιπόν είναι τελευταία φορά που έρχεστε εδώ στην Επιτροπή αυτή ΕΚΟΝ πριν τη λήξη της θητείας της. Τελευταία που θα προεδρεύω εγώ. Περάσαμε αρκετά καλά μαζί όλο αυτό τον καιρό γνωμοδοτήσαμε ε, θετικά για τον ε, ορισμό σας και έκτοτε νιώθουμε κάπως υπεύθυνοι για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η θητεία αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη βέβαια, είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Πριν από λίγο καιρό, ορισμένοι αμφέβαλαν κατά πόσο η Οικονομική και Ένωση θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει. Ευτυχώ και χάρη στι δράσει μεταξύ άλλων και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σήμερα είμαστε μάλλον σε καλή κατάσταση. Βέβαια, ακόμα μένει πάρα πολλή δουλειά να γίνει. Και η γενική αίσθηση είναι ότι θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και εμεί μέχρι το τέλο τη θύρας και επόμενοι τα όσα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συνεργασία τη Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχιστεί, προβλέπεται εξάλλου και από το πακέτο των έξι συμφωνιών και με την Τραπεζική Ένωση επίση, για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Άκουσα σχόλια από κάποιου ότι περνάμε πάρα πολύ καιρό να σε ρωτάμε άλλα πράγματα και όχι για την νομισματική πολιτική στις συναντήσεις μας αυτές. Αλλά με την νομοθεσία που είχαμε και με τις επιπτώσεις επί της νομισματικής ένωσης, νομίζω ότι για όλους μας ήταν καλό που είχαμε την ανταλλαγή απόψεων αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα και ρωτούσαμε και άλλα πράγματα πέρα από τα επιτόκια. Βέβαια και με άλλες κεντρικές ε, τράπεζες αποφασίσατε για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής μας. Στο μέλλον, δίχως άλλο, θα χρειάζεστε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να ξέρετε ότι χαρήκαμε πολύ όσες φορές σας είχαμε εδώ που μας απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, μερικές φορές που δεν ήταν τόσο συνηθισμένες, αλλά και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά νομίζω ότι βοηθήσαμε στο νομοθετικό έργο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ μέλη. Είναι η τελευταία μου ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων πριν από το τέλος της θητείας. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω Σάρων για τον τρόπο με τον οποίο κατήφθηνες εργασία της Επιτροπής ε, μέσα σε μια δύσκολη περίοδο. Όπως είπες, ναι, συνεργαστήκαμε άριστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την ειλικρινή και καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων που διεξήχθη τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ήταν ε, ανεκτήμητη η εμπειρία αυτή για μένα. Δύσκολη καιρή, δύσκολη κρίση και αυτό το θέμα της λογοδοσίας με ευρωπαϊκές προοπτικές ήταν κάτι σημαντικό σαν θέμα για να δεχτεί το κοινό της δράσης μας. Εν γέννη λοιπόν, οι ακροάσεις πάντα ήταν ευπρόσδεκτη ευκαιρία συζητήσεως της οικονομικής καταστάσεω, οικονομικής και ενασματικής ενώσεως μεταξύ δύο πραγματικών ευρωπαϊκών θεσμών και η συζήτηση περί τη σωστή πορεία βοήθησα. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της προσεγγίσεως με μια νέα Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων μετά τον Ιούλιο. Δράτω με της ευκαιρίας της τελευταίας ακροάσεως να κάνω μια αποτίμηση νομισματικής πολιτικής που άσκησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία πενταετία και να αναθεωρήσω τα επιτευχθέντα στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια των ετών αυτών επιτρέψτε μου να προβώ σε μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν υπησέλθω σε λεπτομερή ανάλυση των τριών τομέων, να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας γίνεται, τράπεζα, συγγνώμη, γίνεται την Πέμπτη. Εν όψη λοιπόν της επικειμένης περίοδου προετοιμασίας, αν θέλετε, δεν θα μπορέσω να σας κάνω μια ανάλυση γιατί αναμένουμε την περίοδο Πούρντα όπως αναφέρεται, όπως λέγεται. Την επόμενη πενταετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα περασμένα πέντε χρόνια έλαβε τα αναγκαία μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να διατηρεί σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη. Θέλω να στραφώ στην πρώτη ακρόαση αυτού του κοινοβουλίου, τη θητεία του κοινοβουλίου που έλαβε χώρα με τον προκάτοχό μου το Σεπτέμβριο του 2009 τότε η οικονομία έφτανε στο, στον αδύρ της μετά τη μεγάλη συστολή που ακολούθησε την ε, χρεοκοπία του, της εταιρείας Lehman. Υπήρξαμε μάρτυρες αρνητικού πληθωρισμού. Σε αυτό το περιβάλλον η προοπτική εν γέννη θεωρείται ότι θα με την προσέγγιση για σταθερότητα των τιμών. Ο πληθωρισμός προβλεπόταν να αυξηθεί προς επίπεδα περίπου του 2% το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πάγωσε σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στα επίπεδα εκείνα στα οποία έφτασαν μετά από διάφορα στάδια μετά το φθινόπωρο του προηγουμένου έτους. Κάποια σταδιακή εξάλληψη μη τυπικών μέτρων ε, ανακοινώθηκε. Όμως ε, τον Μάιο του 2010 το κρατικό χρέας και οι αγορές, οι σχετικές πάγωσαν σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης υπήρξε κατακαιρματισμός χρηματοπιστωτικός και έλαβε νέες μορφές άγνωστες με οικονομικές συνθήκες και διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής που πήκυλε από χώρα σε χώρα. Ανταποκριθήκαμε θεσπίζοντας το πρόγραμμα για τις αγορές χρεογράφων εστιαζόμενοι στις αγορές κρατικών ομολόγων. Αρχικά ενώ ο οικονομικός αντίκτυπος των κρατικών χρεών ήταν περιορισμένος εμείς και περιοριζόταν σε ευάλωτες οικονομίες, η ταχεία ανάκτηση σε παγκόσμιο επίπεδο έθεσε πιέσεις επί των τιμών των ενεργειακών. Και αυτό οδήγησε σε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αποφασίσαμε να αυξήσουμε τα επιτόκια αρχές του 2011 βλέποντας ότι θα υπήρχαν κίνδυνοι για τον πληθωρισμό λόγω των τιμών της ενέργειας και λόγω ε, της ρευστότητας της νομισματικής που ήταν μεγάλη. Όμως το κρατικό χρέος επιδεινώθηκε και η Ευρωζώνη μπήκε σε μια δεύτερη ύφεση. Οι πληθωριστικές πιέσεις που εμφανίστηκαν προηγουμένως υποχώρησαν. Γι' αυτό μειώσαμε τα επιτόκια σε μια σειρά σταδιακή με διάφορα βήματα οι πιέσει της αγορές του κρατικού κρέους τελικά υπονόμευσαν ε, την δυνατότητα χρηματοδότησης των τραπεζών σε αυτά τα κράτη-μέλη που είχαν προβλήματα. Για να σταματήσουμε μια συρρήκνωση, μια κατάρρευση όσον αφορά το σωτικό τομέα, δώσαμε, χρηματοδοτήσαμε διάφορες επιχειρήσεις ε, προσπαθώντας να πετύχουμε ρευστότητα σε σταθερό επιτόκιο. Υπήρξε αμοιβαία έκθεση των τραπεζών και των κρατών και τελικά μπήκαμε σε μια κρίση εμπιστοσύνη. Οι επενδυτές λοιπόν ξεκίνησαν, άρχισαν να φοβούνται όσον αφορά ε, τα χρεόγραφα τα, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Θεώρησαν ότι δεν θα μπορούσαν αυτά να πληρωθούν στο δικό μας κοινό νόμισμα. Οπότε υπήρχε κίνδυνος ε, υποτίμησης πάρα πολύ σημαντικός. Όπως ξέρετε η ακεραιότητα της Ευρεζώνης είναι απόλυτη προϋπόθεση για μας να μπορούμε να κινηθούμε σωστά βάσει της εντολής που απορρέει από τις συνθήκες και πιο συγκεκριμένα να εξασφαλίζουμε μια ομαλή εφαρμογή της νομισματικής μας πολιτικής. Για να διατηρήσουμε την εν λόγω ακαιρεότητα ανακοινώσαμε την ετοιμότητά μας να διεξάγουμε άμεσες νομισματικές συναλλαγές ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τους κινδύνους χωρίς να επιβαρύνουμε τα χρεόγραφα. Αυτή η ανακοίνωση αντέστρεψε τις αποσταθεροποιημένες ζωές κεφαλαίων και τους φόβους περί υποτιμήσεως που εμφανίστηκαν την άνοιξη του 2012. Οι χρηματοστικές αγορές ακολουθούσαν σταθερή πορεία προς εξομάλυνση της καταστάσεως και αυτό επί σειρά μηνών. Όμως προς το τέλος της ανοίξεως και αρχές του καλοκαιριού του 2013 οι, νομισματι... οι αγορές χρήματος της Ευρωζώνης όπως και σε άλλα σημεία του κόσμου ε, υπέστησαν εξωτερικούς ε, κλειδονισμούς. Είδαμε ότι αυξανόταν ε, το αναμενόμενο επιτόκιο, το προσδοκόμενο επιτόκιο αυτό ήταν απροσδόκητο εν ώψη των μακροοικονομικών συνθήκων που θεωρούσαμε ότι επικρατούν και δεν τέριαζε με την πολιτική που ήθελε να ακολουθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πέρσι τον Ιούλιο διευκρινίσαμε τους προσανατολισμούς της νομισματικής μας πολιτικής για το μέλλον. Προσφέραμε προσανατολισμό και συμβουλές για το μελλοντικό, μελλοντική πορεία των πολιτικών ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη της σταθερότητας των τιμών. Όλα τα μέτρα μας, τα κανονικά και τα μη τυπικά, τα έκτακτα, ελήφθησαν για να εξυπηρετήσουν το βασικό μας στόχο, δηλαδή σταθερότητα τιμών. Και απέτυχαν τα μέτρα. Από τον Ιούνιο του 2009, δηλαδή από τις αρχές της θητείας αυτής, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ήταν 1,8% σε εξαιρετικές περιστάσεις τα μέτρα μας ήταν εξαιρετικά και αυτά. Όμως και έκτακτα. Αλλά είχαμε βασικό στόχο πάντα. Αμετάβλητο. Η στατικική μας παρέμεινε οδηγός μας. Ήταν φανερό ότι έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό μέσω μακροπρόθεσμα. Βασιζόμαστε στις επιταγές και στους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου. Να παραμείνουν τα επιτόκια κάτω αλλά κοντά στο 2% πρόθεσμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε αποτελεσματική νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να θυμηθούμε ότι πετύχαμε πολλά στον τομέα της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής. Τέσσερα χρόνια μετά που το πρώτο κάτω μέλος ζήτησε οικονομική βοήθεια, σήμερα μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά ότι έχουμε αφήσει τα χειρότερα πίσω μας. Έχουν περάσει. Τα αποφύγαμε. Η πολιτική βούληση όλων των εμπλεκομένων φορέων ήταν αρκετά ισχυρή για να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ. Πολλοί είχαν υποτιμήσει αυτή την πολιτική βούληση. Και η ζωφερή εικόνα που είχε σχηματιστεί όσον αφορά το χρέο και εξακολουθούν να προσπαθούν, παρόλα αυτά η Ευρωζώνη όσον αφορά τα βασικά στοιχεία τα οικονομικά και όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν στις ε, αρχές ε, της εντολής του Κοινοβουλίου, της θητείας του Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι κινούμεθα προς σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να πούμε ότι το ποτήρι είναι τουλάχιστον μισογεμάτο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στη διόρθωση των οικονομικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Οι ανισορροπίες υποχωρούν και τίθενται τα θεμέλια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αυτό αληθεύει όλους ιδίω για χώρες προγραμμάτων που καταβάλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά τους να διορθώσουν τον οικονομικό τομέα, το χρηματοδοτικό, και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομικές τους ε, δομές. Πέρα από τις εθνικές πολιτικές, η Ευρωζώνη έγινε πιο ανθεκτική. Σε, αυτές, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια όπου υπήρχε ο πειρασμός να επιστρέψει κανείς εθνικά μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πραγματικά ευρωπαϊκή προπτική έπαιξε κρίσιμο ρόλο. Εξασφάλισε εφαρμογή πραγματικά ευρωπαϊκών λύσεων. Γνωρίζω ότι η θεσμική προσέγγιση που έπρεπε να ακολουθηθεί σε κάποιες φάσεις δημιούργησε κάποια δυσαρέσκεια, ε, κυρίως στο Κοινοβούλιο. Εν γέννη όμως αναγνωρίζονται τα επιτευχθέντα. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε το, τη δέσμη των 6 μέτρων, των 2 μέτρων και τη, το δημοσιονομικό σύμφωνο Οπότε μπορούσαμε να ανταποκριθούμε με όλα αυτά καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Νομισματική Ένωση. Ήταν σημαντικό βήμα αυτό για ορθά δημοσιονομικά στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, βελτίωση του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό δείχνεται από το CRD4 και από το συμβιβασμό που καταλήξαμε όσον αφορά το BRRD και σταδιακά βήματα που έγιναν προς τα πραγματική τραπεζική ένωση με ενίο υποπτικό φορέα, ενίο μηχανισμό εξυγίανσης και εναρμονισμένο πλαίσιο για διάφορα σχήματα εθνικά για εγγύηση των καταθέσεων. Όλα αυτά θα μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους από μια κρίση παρόμοια με αυτή που περάσαμε. Και μειώνει και την πιθανότητα να επανεμφανιστεί με τέτοια κρίση τέτοιου μεγέθους. Τρίτον, το 2010 δεν υπήρχαν μέτρα και διευθυντήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος των κρατών μελών όταν έχαναν την πρόσβαση στις αγορές. Αυτή η έλλειψη ε, δημιουργούσε μεγαλύτερη βεβαιότητα στις αγορές για τις ενδεχόμενες διεξόδους. Με τον ενίο αυτό μηχανισμό επίλυση ε, των, προβλημάτων και με το, ε, τη δέσμη των διπλών, το 2-pack, με τα δύο μέτρα, ε, βρήκαμε μία διέξοδο, σημαντικό βήμα πρόοδου και στο μέλλον η Ευρωζώνη θα είναι καλύτερα ετοιμασμένη το τρόπος για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κρίσεις. Αν το δούμε ιστορικά το θέμα. Πέντε χρόνια είναι ένα ανοιγό κλίμα του ματιού μόνο. Ένας βλεφαρισμός. Τα τελευταία πέντε χρόνια έκανε τεράστια βήματα πρόοδου η Ευρωζώνη και έτσι μείναμε ενωμένοι. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε να το τονίσουμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι σίγουρος ότι από τον Ιούλιο και πέρα, στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου, θα συνεχίσει να παίζει το σημαντικό ρόλο του, τον ίδιο που έπαιξε και στην προηγούμενη θητεία. Έχουμε προκλήσεις ακόμα μπροστά μας. Είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές, πολύ περίπλοκες δεν μπορούμε να φυσικάζουμε. Είναι πολύ νωρίς να πούμε και να ισχυριστούμε ότι έχουμε εκπληρώσει την αποστολή μας. Οι λαοί της Ευρωζώνης υποφέρουν από τις αναπόφευτες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν μετά από χρόνια συσσόρευσης ανισορροπιών. Η ανεργία παραμένει απαράδεκτα υψηλή. Οι πολίτες κρίνουν την Ευρώπη βάσει της δυνατότητας να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη. Τα επόμενα έτη πρέπει να δημιουργήσουμε πιο τέλεια ένωση που φροντίζει να καλύψει τους προαναφερθέντες στόχους. Πάνω απ' όλα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις αναληφθήσεις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, να διορθώσουν τις ανισορροπίες και να μεταρρυθμίσουν την δομή των οικονομιών τους. Οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να αφιγραμμιστούν με τις διατάξεις του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας και τις διατάξεις της, ε, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Η εξυγίανση, η δημοσιονομική θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη, να είναι φιλική στην ανάπτυξη. Οι διαθετικές αλλαγές θα τονώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο αυτά που σε αντιμετώπισαν σε κάποια φάση την Άβυσο διότι έχασαν την πρόσβαση στις αγορές είναι κάτι που αφορά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού ομοιόμορφα κοινοί κανόνες. Η ανταπόκριση σε ανηληφθήσεις υποχρεώσεις σημαίνει τήρηση υποσχέσεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υποσχέσεις που έγιναν τον Ιούνιο του 2013 σχετικά με την ολοκλήρωση Ευρωπαϊκής Τραπεζική Ένωσης σημαίνει ταχεία ενσωμάτωση οδηγιών σε εθνικό δίκαιο και αυστηρή εφαρμογή του υιοθετηθέντος νομοθετικού ρυθμιστικού πλαισίου. Σημαίνει ότι ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, ο νέος μηχανισμός εξυγίανσης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συμφωνήσουμε πριν από το τέλος της θητείας. Η δημιουργία μιας πιο τέλεια ένωσης απαιτεί την κάλυψη των κενών της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ενώσεως. Χρειάζεται πραγματική συνολική οικονομική και νομισματική ένωση και ε, είναι κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση των τεσσάρων πρόεδρων και εξακολουθεί να παραμένει ύψιστο στόχος μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθούμε στο μέγιστο δυνατόν την ολοκλήρωση. Δεν είναι οικονομικός αναγκαίο, ούτε πολιτικός ε, ρεαλιστικό σημαίνει την ευθυγράμμιση οικονομικής διακυβερνήσεως και των πολιτικών των κρατών μελών, όπου αυτό ενδείκνεται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται να ε, τονίζουμε τα θετικά αποτελέσματα και να εξουδετερώνουμε τις εξωτερικές αρνητικές πιέσεις. Χρειάζεται ένας επιμερισμός της κυριαρχίας σε κρίσιμους τομείς. Αυτή είναι μία λύση, είναι μία προσέγγιση για την επίτευξη των παραφερθέντων στόχων. Η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να ε, διατάξει λύσεις. Αυτό είναι ένα πολιτικό προνόμιο. Και ελπίζω και σαν υπεύθυνο για Τράπεζα και σαν Ευρωπαίος πολίτης ότι η επικείμενη προεκλογική εκστρατεία θα είναι μια ευκαιρία ούτω ώστε να διεξαχθεί μια συζήτηση επιλύσεων για τον κοινό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον η Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στις ερωτήσεις. Thank you. Uh, we will go straight Ευχαριστώ. Πάμε σε ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτα για το ΕΛΚ. Ε, κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς. Κύριε... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μέχρι να βρει ο ο ναι. κύριος στο σωστό κανάλι. Επαναλαμβάνω ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις δηλώσεις σας και ιδίως για τον έπαινο που απευθύνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο του προερχόμενος από την Γερμανία γνωρίζω ότι υπάρχουν και θεσμοί που δεν το κρίνουν έτσι το πράγμα και αυτό σας ευχαριστώ. Πρώτα για το ίδιο κεφάλαιο σε κρατικά δάνεια. Εδώ και καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί κάποιες αλλαγές. Στις διαπραγματεύσεις με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνδέονται, μάλλον απορρίπτεται η σύνδεση των κρατικών δανείων με τον ίδιο κίνδυνο. Και πρόσφατα μάλιστα και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το ίδιο. Γι' αυτό και ρωτώ κύριε Πρόεδρε εσείς ποια άποψη έχετε και κυρίως όσον αφορά την ανάγκη να γίνουν κάποια πρώτα βήματα κυρίως εν ώψη των στρέστες, των δοκιμασιών αλλά και για πιο μακροπρόθεσμα μέτρα. Δεύτερο, για την Τρόικα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στην Τρόικα στις ε, χώρες όπου σημειώνουν τα προβλήματα και όπου δραστηριοποιείται η Τρόικα σημειώνεται κριτική για τα μέτρα εφαρμογής παρόλο που τα μέτρα και συχνά και, η εθνική τα εθνικά κοινοβούλια έχουν συνδιαπραγματευτεί. Δείχνει όμως η πρόσφατη εμπειρία ότι οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει από την ε, θεραπεία εντό εικόνα αυτή, πολύ σύντομα μετά από λίγα χρόνια δηλαδή, ανακάμπτουν. Τι γνώμη έχετε εσείς. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σημείο, για τη στάθμιση του κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα, πρέπει να κάνουμε με διάκριση. Πρέπει να διακρίνουμε τι διάφορε στοιχέ. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η γενική στάθμιση των κρατικών ομολόγων συναρτήσει των αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και στις ρυθμίσεις που αφορούν, αφορούν τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας και θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις τράπεζες στον κόσμο. Υπό τη μορφή ενός παγκοσμίου κανονισμού. Άλλη πτυχή. Ποια θα είναι η αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων στην αναθεώρησή μας όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού Εκεί η αξιολόγηση θα ακολουθήσει το τρέχον CRD4 και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τρίτη πτυχή. Αυτά τα κρατικά ομόλογα πώς θα αντιμετωπιστούν στις δοκιμές αντοχής, stress test, απάντηση. Όπως και όλα τα άλλα στοιχεία ενεργητικού θα υποστούν δοκιμασία αντοχή σύμφωνα με τις ε, παραμέτρους αντοχής όπως και τα άλλα στοιχεία ενεργητικού. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συντηρητικοί τώρα, δοθήσεως της καταστάσεως του παρόντος κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του πλαισίου που υπάρχει. Δεύτερο ερώτημα, η Τρόικα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι χώρες που εντάχθηκαν στα προγράμματα στα οποία κινητοποιήθηκε η Τρόικα, ωφελήθηκαν από αυτές τις διαδικασίες, αυτά τα προγράμματα. Μπορούμε να τα πούμε ε, τώρα έχοντας χρόνια πίσω μας δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, ο δρόμος ήταν δυσκολότατος, πάρα πολύ οδυνηρό στις περισσότερες ε, περιπτώσεις, όμως είναι σαφές ότι αυτά τα προγράμματα σε μεγάλο ποσοστό ήταν αυτό που χρειαζόταν και χρειάζονται αυτές οι χώρες διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο μας. Ίσως για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα θα έχω τη δυνατότητα να το εκθέσω αυτό το θέμα. Το βασικό στοιχείο ποιο είναι ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα είχε στόχο τη βελτίωση της επιβολής των νομισματικών μας πολιτικών. Πρώτιστα, να έχουμε καλύτερη διέξοδο, δίευλο για τις νομισματικές μας πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ελίζα Φεραίρα τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Αγγλικά θα μιλήσω για να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, λέει η κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν, στη θέση που ήσασταν όταν έφτασε η κρίση. Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο μου για να τα επαναλάβω όλα αυτά, θέλω όμως να σας ρωτήσω, μάλλον να σας ζητήσω, να μην σταματήσετε να σκέφτεστε και να προτείνετε τι λείπει από το αρχιτεκτόνημα αυτό της Ευρωζώνης. Ξέρω θα το κάνετε, αλλά θέλω να επικεντρωθείτε σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας ε, για τον μηχανισμό εξυγένσης. Ξέρετε ότι είναι κάτι που βέβαια συνδέεται άμεσα με τις τράπεζες και νομίζω ότι βοήθησε και στην περίπτωση του SSM, του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Είμαστε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις τώρα με το Συμβούλιο. Ως εισηγήτρια λοιπόν και στο όνομα της ομάδας, ε, εισηγητή, σχεδόν εισηγητών, συνεισηγητών κτλ. Θέλουμε να σας ζητήσουμε να είσαστε ξεκάθαρος στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διαδικασία αυτή. Γιατί έχετε την νομιμότητα να το κάνετε, επειδή η δικιά σας η εποπτεία δεν θα είναι αξιόπιστη αν συγχρόνως δεν έχετε και ένα ισχυρό πλαίσιο εξυγίανσης τραπεζών. Πρέπει να είναι μια διαδικασία που δεν περνάει από την πολιτικοποίηση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση μετά τις διαδικασίες ε, διάσωσης. Το άλλο που θέλω να ζητήσω είναι το εξή. Όταν έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα στις διάφορες χώρες, εντάξει εδώ δεν θέλω να σχολιάσω τα θετικά σας σχόλια, ξέρετε ότι που συμφωνούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί. Ορισμένες χώρες βγαίνουν από πρόγραμμα με 30-50% υψηλότερο δημόσιο χρέος. Δεν υπάρχουν αρκετές προοπτικές ανάπτυξης ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος αυτό, οπότε ρωτάω η ανακοίνωση για το MT εξακολουθεί να ισχύει. Θα μπορέσετε να παρέμβετε εάν χρειαστεί για την αγορά δηλαδή ε, δημοσίων ομολόγων και χρέους για να προστατεύσετε τις χώρες από νέες κερδοσκοπικές τάσεις. Ευχαριστώ. Απάντηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να καταλήξουμε σε ένα καλό συμπέρασμα όσον αφορά τον ΙΣΕΡΕΜ. Η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η δικιά μου είναι σαφής από την αρχή που έχει, γίνει, που έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Λέμε το ίδιο ότι λέγαμε και στην αρχή, ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να έχει μια αποτελεσματική διακυβέρνηση και κατάλληλη, ικανή να παίρνει αποφάσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες πολλές φορές και αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται επίσης και γρήγορα χωρίς ε, προβλήματα και συγκρούσεις. Δεύτερον, πρέπει επίσης να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αξιολόγηση που κάνει η SSM, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Υποπτική Αρχή δηλαδή, και οι αποφάσεις που παίρνονται από τον ESRM. Ο ενίος υποπτικός μηχανισμός θα αξιολογεί κατά πόσο μια τράπεζα πρέπει ή όχι να εκαθαριστεί ή, για να το πω καλύτερα, δεν είναι βιώσιμη από μόνη της πια και ο ESRM θα αποφασίζει τι είδους, πώς θα γίνει αυτή η εκαθάριση και θα παίρνει τις αποφάσεις μετά την αξιολόγηση του εποπτικού μηχανισμού. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο, είναι διακριτά. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι καλό, μεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΡΕΜ, αλλά ως παρατηρητές θα είμαστε εκεί. Το τρίτο σημείο. Πόσος ο χρόνος χρειάζεται, 10 χρόνια έχουμε πρα, πριν υπάρξει ένας κοινό μηχανισμός ώστε οι κίνδυνοι να αμοιβεοποιούνται, να είναι κοινοί. Είπαμε ότι χρειάζεται πολύ χρόνος. Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα, αυτό εξάλλου δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες θα καλούνται να πληρώνουν δύο φορές πιο γρήγορα, αλλά θα σημαίνει αν μη τι άλλο ότι θα υπάρχει κάτι κοινό μετά τη μεταβατική πρώτη περίοδο των 5 ετών. Και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτή, αυτό το κοινό backstop σημαίνει ότι η SRM θα μπορούσε να δίνει εγγύσεις ή θα μπορούσε να υπάρχει μια πιστοτική γραμμή στον ESRM. Για μας αυτά είναι τα στοιχεία κλειδί για τον μηχανισμό αυτό. Εγώ δεν λέω ότι ο νέος εποπτικός μηχανισμός δεν θα είναι έτοιμος και δεν θα μπορεί να κινητοποιηθεί. Αλλά αν ο Ιασαρέμ δεν υπάρχει, τότε υπάρχει μπέρδεμα αρμοδιοτήτων. Θα έχετε ένα κεντρικό σώμα το οποίο θα παίρνει μια απόφαση και μετά θα είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες θα αποφασίζουν για την εκαθάριση. Άρα εκεί μπορεί να υπάρξει μπέρδεμα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες. Τώρα για το OMT, το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Είναι έτοιμο και μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Αρχίζει και με όλες τις ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στο σχεδιασμό του μηχανισμού αυτού. Είναι ένα πρόγραμμα μια συγκεκριμένης φύσης και ενεργοποιείται κάποιες συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτού. Ευχαριστώ. Παρέβασε εκτός μικροφώνου για την Τρόικα. Δεν μου είπατε για την Τρόικα. Καμία σχέση. Με ρωτήσατε για το MT, Outright Monetary Transaction, αγορά χρέους. Σας απάντησα. Πρόεδρος. Έτσι κι αλλιώς, αν με την ερώτησή σας φάτε πάνω από το μισό χρόνο σας, εννοείται ότι η απάντηση δεν θα είναι πλήρης. Εκ μέρους του Άλντε τώρα, Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η τελευταία φορά που θα έχω την ευκαιρία να σας υποβάλω ερωτήσεις και προσωπικά για αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου και το θαυμασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο ε, διαχειριστήκατε την κρίση σαν διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας. Πολλοί συνάδελφοι θα πούν αυτό, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω μια και είναι η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο. Έχω δύο ερωτήσει. Για την Ουκρανία, πρώτα απ' όλα. Είναι στο μυαλό όλων η Ουκρανία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να σχολιάσετε το θέμα. Και πώς οι προσδοκίες για την Ευρώπη επηρεάζουν διαμόρφωση νομισματική σας πολιτική. Η ερώτησή μου λοιπόν, διαφάνεια. Είπατε ότι έχουμε πέντε χρόνια μπροστά μας. Έχουν περάσει πέντε χρόνια μάλλον. Και ο έλεγχος και η διαφάνεια θα μπορούσαν στο μέλλον να βελτιωθούν. Θα προσπαθήσετε να δημοσιεύετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων σας την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, η διχασμένη Ευρώπη. Προέρχομαι από χώρα εκτός Ευρωζώνης. Πάντα υποστήριζα το ευρώ και στο να προσχωρήσει η χώρα μου στο ευρώ. Μιλήσατε για μια τέλεια ένωση. Δεν θα είναι διχασμένη η Ευρώπη έτσι που θα διαμορφωθεί με την Τραπεζική Ένωση και τα άλλα μέτρα που εστιάζονται επί των χωρών της Ευρωζώνης. Φοβάμαι ότι με αυτά τα μέτρα τελικά θα έχουμε μια διχασμένη ε, Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Δράγκη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και τα συγχαρητήρια γιατί αυτά είναι αγαθά ε, που σπανίζουν και γι' αυτό τα χαίρομαι και ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Όμως δεν κατάλαβα καλά τι εννοείται για την Ουκρανία. Θέλετε να σχολιάσω την κατάσταση στην Ουκρανία. Εδώ υπάρχουν βέβαια περίπλοκες απαντήσεις. Μπορεί κανείς να δώσει μια απάντηση δυσδιάστατη. Αφενός καθαρά τεχνική, οικονομική διάσταση, αλλά θα έλεγα πιο στενή οικονομική διάσταση και εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρέπει να εξετάσουμε τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς της Ουκρανίας με την ζώνη ευρώ και είναι μάλλον περιορισμένοι. Είναι λιγότερο από 1% των ευρωπαϊκών εξαγωγών, μάλλον της ζώνης ευρώ και λιγότερο από 1% των ε, ε, αξιώσεων των Ευρωπαϊκών Τραπεζών είναι απέναντι σε αντισυμβαλόμενους από την Ουκρανική πλευρά. Συνολικά λοιπόν από την άποψη, από τη στενή αυτή η οικονομική άποψη, η επίπτωση στη ζώνη ευρώ θα είναι πιθανότατα σχετικά περιορισμένη. Πάλι εδώ θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με τα όσα συνέβησαν όχι εδώ, ε, εδώ και όχι πολύ καιρό από τις ε, οικονομικές αποφάσεις που λήφθηκαν από άλλες χώρες και είδαμε ότι η επίπτωσή τους στην ε, ζώνη ευρώ ήταν περιορισμένη. Όμως η γεωπολιτική διάσταση της κατάστασης όπως διαγράφεται εκεί είναι βεβαίως μια πολύ διαφορετική ιστορία όπως είδαμε και από τα spillover ε, των αναφιόμενων αγορών. Και οι γεωπολιτικές διαστάσεις της ε, καταστάσεως αυτής μπορούν οι ίδιες να αναπτύξουν μια δύναμη και ένα δυναμικό επιρροής σε γεγονότα που ίσως να είναι πολύ πέραν των στατιστικών αριθμών που μόλις σας ανέφερα προηγουμένως. πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση ιδιαίτερα προσεκτικά και γνωρίζοντας ότι δεν είναι μοναχά θέμα λήψης αποφάσεων οικονομικής πολιτικής, αλλά το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και ίσως να έχει επίπτωση και στην οικονομία. Για την διαφάνεια τώρα, το θέμα που θίξατε και για τα πρακτικά, αρχίσαμε όπως είχε προταθεί προκαιρού. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο μια πρόταση για τη δημοσίευση των πρακτικών. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα πρώτο γύρο συζητήσεων. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Έχω πει και άλλη φορά, με άλλη ευκαιρία, ότι η συζήτηση αυτή είναι περίπλοκη, γιατί καλούμαστε να εξετάσουμε διάφορες πτυχές γιατί πρέπει να είναι και ενημερωτικά και διαφανή. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορώ όμως να σας βεβαιώσω ότι η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί πριν από την πάροδο της πενταετίας και ότι θα δημοσιευθούν τα πρακτικά πριν να περάσουν τα πέντε χρόνια. Νομίζω ότι μπορώ να σας το υποσχεθώ αυτό. Θέσατε και ένα άλλο θέμα. Όντως πολύ παρόν στο πνεύμα μας. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για την Τραπεζική Ένωση προκαλούν και διαστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για τα φυσιολογικά βήματα που πρέπει να λάβει η Νομισματική Ένωση για την αυτοσυντήρησή της. Η Νομισματική Ένωση ήδη απετέλεσε ένα τολμηρό βήμα προς τα ευρώ, είναι όμως ατελής. Υπάρχουν πλείονα βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμη πριν να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι η αρχιτεκτονική της νομισματικής ενώσεως είναι πλέον στέρεα. Ένα από τα βήματα αυτά είναι και η Τραπεζική Ένωση. Θα υπάρξουν και άλλα βήματα Το ερώτημα είναι τι γίνεται με όσους δεν συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ. Η Τραπεζική Ένωση, ως τώρα τουλάχιστον, έχει εμφανιστεί ως ανοιχτός σχεδιασμός. Δηλαδή, όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα μπορέσουν να το πράξουν. Έχουμε και διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του SSM μας, η SP, και των εποπτικών αρχών χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη. Αλλά όπως είπα είναι ανοιχτός σχεδιασμός, άρα δεν είναι αποκλειστικό όργανο, αποκλειστική λέση. Ευχαριστώ. Προσπαθήστε να ρωτάτε λιγότερες ερωτήσεις, αλλιώς θα βρεθούμε σε δυσκολία. Έπινγκ. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, το 2012 είπατε ό,τι και αν χρειαστεί. Οπότε ξαφνικά μετατραπήκατε σε James Bond του νομισματικού κόσμου έχετε και άδεια να τυπώσετε. Λοιπόν, αυτό ε, για την ώρα με το πρόγραμμά σας έχει φυσικάσει ο κόσμος της οικονομικής αγοράς, αλλά το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας σας δημιούργησε προβλήματα. Λοιπόν, πιστεύει ότι το MT είναι κάτι παράνομο και ασύμβατο με το γερμανικό δίκαιο και εφόσον το δικαστήριο έχει μόνο δικαιοδοσία για γερμανικό δίκαιο παρέπεμψε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι ο κ. Γκάουάιντερ της Bundestag από το ίδιο κόμμα τον κύριο Φέρμπερ θα τρέξουν στην κασλούη για να α, αντισταχθούν στην συμμετοχή της Bundesbank στο OMT. Άρα η άδειά σα μέχρι να τυπώνετε, μέχρι ποιο σημείο φτάνετε. Και η αντίδραση γερμανική δεν δείχνει ότι είσαστε εκτός, μάλλον δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι χρειαστεί όπως είχατε δηλώσει, σαν James Bond με άλλα λόγια. Κατά τη γνώμη μας οι OMT είναι απολύτω νόμιμοι και εμπίπτουν στο πλαίσιο τη εντολή μα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ναι, ναι. διαθέτει αυτή την εντολή. Τώρα το ότι θα κάνει η Bundesbank ή όχι θα πρέπει να του ρωτήσετε του ίδιου. Χωρί να λησμονείτε όμω την κατανομή του κινδύνου, το risk sharing και αυτό λέχθηκε στο ακροατήριο στην Καλσρούη. Διότι αυτό επιβαρύνει όλου είτε συμμετέχουν είτε όχι. Ευχαριστώ δεν Με άλλα λόγια, ε, κανείς έχει το όπλο στην τσέπη του, δεν σημαίνει ότι πυροβολεί κιόλα. Γκίγκολτ, για τους πράσινους. Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση που αφορά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις αγορές. Και εσείς, από ό,τι θυμάμαι, και οι προκάτοχοί σας ήταν υπερήφανοι, πολύ περήφανοι, ότι παρά τα σκαμπανεβάσματα, βραχυπρόθεσμα, ε, μακροπρόθεσμα μάλλον ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στο, κοντά στο 2%. Υπάρχει διακύμανση των αγορών. Από 1,5 μέχρι 1,7 αν το πάρουμε σε διάρκεια δεκαετίας δεν είναι κοντά στο 2%. Πώς το βλέπετε εσείς, ποιες είναι οι συνέπειες αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό ή την νομισματική της πολιτική. Θα θέλαμε λεπτομέρειες. Αυτά τα γεγονότα πώς επηρεάζουν την προσέγγισή σας. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να είσαστε υπερήφανος όπως κατά το παρελθόν ότι επιτυγχάνετε τους στόχους σας πλήρως. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις τιμές, να, δεν θα πρέπει ποτέ να είμαστε να αισθανόμαστε υπερηφάνεια ενώ πρόκειται για συλλογικές προσπάθειες πολλών εκατομμυρίων υποκειμένων. Αυτό που μπορούμε να πούμε, καθώς στρέφουμε τα βλέμματα προς τα πίσω, να το πούμε κάποια ικανοποίηση, βλέποντας ότι λίγο πολύ τα τελευταία 15 χρόνια η, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέδωσε, οι προσπάθειες της απέδωσαν και αν κάνετε και συγκρίσεις και με άλλες τράπεζες αλλού, ακόμα και πριν να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δείτε λοιπόν ότι το ιστορικό της είναι, είναι το ιστορικό είναι ικανοποιητικό, αλλά αρκούμε στο ικανοποιητικό, όχι παραπάνω. Για τον προσδοκόμενο πληθωρισμό ή τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Εξακολουθούμε να θεωρούμε τον μέσο αναμενόμενο πληθωρισμό να κινείται γύρω στα 2%. Αλλά, αλλά, μια στιγμή. Έχουμε τώρα ένα επίπεδο πληθωρισμού που είναι ασφαλώς χαμηλότερο από το 2%. Αρκετά χαμηλότερο. Και το βλέπουμε αυτό για ένα μεγάλο ε, χρονικό διάστημα, όχι τόσο σύντομο. Πρώτο λοιπόν γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερο παραμείνει ο πληθωρισμός στο επίπεδο αυτό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι ο κίνδυνος να μην επιστρέψει στο 2% εύλογα. Δηλαδή τόσο μεγαλύτερο θα είναι ο κίνδυνος, ο αναμενό πληθωρισμός να ξεφύγει. Και αυτό δεν το θέλουμε. Το δεύτερο, εάν πούμε ότι κάποια στιγμή ο πληθωρισμός θα ανέλθει προς το 2% έστω και μετά από μακρόχρονικο διάστημα, σχετικά μακρόχρονικο διάστημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί. Δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα πιέσουν τον πληθωρισμό να επανέλθει στο 2%. Και εδώ πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε ποιες είναι οι πηγές και οι αιτίες των χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού. Πρώτα υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια διάσταση των χαμηλών τιμών ενεργείας και τιμών τροφίμων. Και αν συγκρίνεται τον, το δικό μας ποσοστό πληθωρισμού με το αμερικανικό θα δείτε ότι των ΗΠΑ δεν είναι και πολύ υψηλότερο, παρόλο που η ανάκαμψή του είναι πολύ πιο προχωρημένη από ό,τι στη δική μα περίπτωση. Επίση, εάν επανέλθουμε στον ρυθμό του πληθωρισμού μετά από την ασιατική κρίση, στα τέλη τη δεκαετία του 90 και μετά την κρίση τη Lehman Brothers το 2009, πάλι θα περίπου τα ίδια. Άρα δεν είναι άνευ προηγουμένου. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε. Εάν αφαιρέσετε την παράμετρο ενέργειας και τροφίμων και εντοπίσετε τον πυρήνα του πληθωρισμού, θα δείτε ότι η πτώση του πυρήνα του πληθωρισμού οφείλεται στην προσαρμογή που έγινε στις τέσσερις ε, χώρες του προγράμματος, των ε, ενισχύσεων, της ενισχύσεως δηλαδή, το, κατά το μεγαλύτερο μέρος λόγω της προσαρμογής των τιμών. Αν όντως είναι έτσι, τότε γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας παράγοντας εφάπαξ. Αφού θα γίνει λοιπόν αυτή η προσαρμογή, τότε ο πληθωρισμός θα αρχίσει πάλι να ανέρχεται. Και εδώ σας περιγράφω τώρα όλη την περιπλοκότητα της αναλύσεώς μας, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και την άλλη πλευρά της ιστορίας δεν είναι μονάχα η πλευρά της προσφοράς είναι και της ζήτησης και θα δούμε ότι με τόσο υψηλή ανεργία η ζήτηση θα παραμείνει ασθενής για κάποιο διάστημα. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και αυτόν τον παράγοντα και να δούμε ότι η μείωση της ανεργίας και εάν περάσει η ανάκαμψη από τον τομέα των εξαγωγών στον εγχώριο τομέα, επίσης αυτό θα είναι πολύ σημαντικό ως παράγοντας. Και εδώ να προσθέσω κάτι ακόμη. Σχετικά και με ορισμένες παρατηρήσεις που έκανα για τον πληθωρισμό. Να συνεχίσω ή να διακόψω εδώ. Α, μπορώ να συνεχίσω. Η σχετική προσαρμογή τιμών γίνεται κυρίως στους τομείς που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό, για παράδειγμα εξαγωγές. το υπόλοιπο της οικονομίας πρέπει να προσαρμοστεί και αυτό. Γιατί αλλιώς θα έχετε χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερους πραγματικούς μισθούς στον προστατευόμενο τομέα. Και όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο δυσκολότερη θα είναι η συνολική προσαρμογή της οικονομίας. Και γι' αυτό χρειάζεστε, και γι' αυτό επιμένουμε πάντοτε ότι χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί εκεί οι αλλαγές θα παίξουν, σε αυτούς τους τομείς θα παίξουν οι αλλαγές ένα ρόλο, δηλαδή στους τομείς που είναι προστατευμένοι από τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για να δούμε τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Κυρία Ματάου. Ματίας. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ μια ερώτηση, ερώτηση όμως που δεν ακούστηκε μέχρι τώρα από τους συναδέρφους και που έχει να κάνει με το πρόβλημα της ρευστότητας, ένα ενδογενές πρόβλημα και που δεν θα το λύσουμε μειώνοντας τα επιτόκια. Ακούμε διάφορα νέα που έχουν να κάνουν με μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτό το τομέα και μία από τις ιδέες που έχει προταθεί είναι να υπάρχει αρεσιμότητα τη στιγμή που γίνεται ανακεφαλοποίηση μια τράπεζας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν προϋποθέσεις που θα έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων για μια τράπεζα προκειμένου να προχωρήσει αυτό. Θέλω να μου πείτε, όντως είναι κάτι που το προβλέπετε εγώ συμφωνώ. Απλώς λυπάμαι που η πρόταση αυτή έρχεται έξι χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης από την οποία όλοι υποφέρουμε. Και λυπάμαι λοιπόν που έξι μήνες μετά την κρίση έχουμε μια τέτοια ε, πρόταση. Βέβαια καλή αργά παρά ποτέ. Τώρα σε τι πλαίσια θα επιβληθεί η ρεσιμότητα αυτή σε αύξηση πιστώσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή τι, ποια θα είναι η προϋπόθεση, πώς ε, θα βελτιωθεί η οικονομία. Ε, Καταπολέμηση της ύφεσης, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όπου με τις αλλαγές στην νομισματική μας πολιτική και τα επιτόκια θα ανταποκρινόμαστε στην κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Θέλω να πω εδώ ότι έχουμε δει πολύ σημαντική πρόοδο από τον Ιούλιο του 2012 όταν ο Τζέμις Μπόντ είπε αυτά που είπε. Έγινε. Για τη χρηματοδότηση έχει πάψει ο κατακαιρματισμός των τραπεζών. Αν δείτε τη βάση καταθέσεων για τις τράπεζες, θα δείτε ότι είμαστε στα ίδια επίπεδο όπως ήμασταν το 2007, οπότε ο κατακαιρματισμός αυτός από τις καταθέσεις έχει σταματήσει. Υπάρχουν μεγάλες βελτιώσεις και στην έκδοση ομολόγων κλπ. Από πλευρά δανεισμού εδώ η πρόοδος είναι πολύ λιγότερη. Αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια πρόοδο και εδώ. Βλέπουμε ρευστότητα χαμηλή μεν, αλλά βλέπουμε να υπάρχει, βλέπουμε και από τις έρευνε που έχουμε κάνει για το δανεισμό των τραπεζών, βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόοδος και σε αυτό το μέτωπο χαμηλή μεν, αλλά το βασικό εδώ, αυτό που είναι ζωτική σημασίας, είναι ότι προκειμένου να υπάρξει αύξηση του δανεισμού χρειάζονται δύο πράγματα. Από την προσφορά, πρώτα απ' όλα, πρέπει η αντίληψη κινδύνου από τις τράπεζες να μειωθεί. Μέχρι τώρα οι χώρες με τη μεγάλη κρίση ήταν χώρες με τη μεγαλύτερη ύφεση, οπότε ο δανεισμός βέβαια ήταν πιο επικίνδυνος από ότι ήταν αλλιώς. Συνεπώς αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί για την προσφορά του δανεισμού. Υπάρχει όμως και το θέμα της ζήτησης για να υπάρχουν περισσότερες πιστώσεις χρειάζεται να υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζητούν πιστώσεις και ζητούν πιστώσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν έχουν πελάτες για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Σε μία από τις έρευνες που έγινε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 8-9 μήνες ρωτήθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δυσκολεύεστε για να προχωρήσετε με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Και η απάντηση, η πρώτη απάντηση ήταν δεν έχουμε πελάτες. Και η δεύτερη απάντηση ήταν δεν έχουμε πιστώσεις. Το δεύτερο δηλαδή που τους απασχολούσε. Άρα από πλευράς των τραπεζών όντω βλέπουμε ότι δυσκολεύονται οι τράπεζες να δώσουν δάνεια, δεν δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που δεν έχουν πελάτες. Οπότε δυστυχώς η εικόνα είναι αυτή που είναι. Έχει βελτιωθεί βέβαια πολύ τον τελευταίο καιρό. Βλέπουμε καλύτερη κατάσταση και από τις ερευνές μας και σε ένα βαθμό και από τα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά τις πιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποια μικρή βελτίωση. Τώρα, τη σχέση συνδέσατε εσείς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το δανεισμό, με τα προγράμματα δανεισμού. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα μέσα που έχουμε, ένα από τα εργαλεία που έχουμε στον ε, ξοπλισμό μας, τόσο πάντων να μην τον πω στον κατάλογό μας, στη λίστα μας. Και προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό, το σκεφτόμαστε. Έχει πολλά όπλα εδώ μαζί του. Τώρα εκ μέρους του EFD, Σάμπο Τέρχο. Ευχαριστώ. Θα υποβάλω την ερώτησή μου στα φιλανδικά. Ε, κύριε Ντράγκη, σας ευχαριστώ που ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Επιτροπή μας και στην ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να συνεχίσω με ένα θέμα που ανέφεραν οι δύο προλαλήσαντες. Εγώ έχω κάπως διαφορετική άποψη. Όπως είπατε στην παρέμβασή σας, βασικός στόχος της ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας ήταν η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Και σύμφωνα με κάποιους έχει πετύχει, σύμφωνα με κάποιους άλλους έχει πετύχει υπερβολικά καλά. Εγώ είμαι από τη Φινλανδία σε σύγκριση με τη Σουηδία η κατάσταση είναι ιδιαίτερη. Πολλοί πιστεύουν ότι η ανταγωνιστικότητα της Φιλανδίας υποφέρει λόγω ισχυρού ευρώ, εν συγκρίση με τη Σουηδία παραδείγματο χάρη. Βέβαια το θέμα είναι πολύ ευρύτερο, δεν αφορά μόνο δύο σκανδιναβικές χώρες, αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης και πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πολλοί διαμαρτύρονται και θεωρούν ότι είναι πολύ ισχυρό το ευρώ. Θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπαν οι πράσινοι. Α, αυτή την ανησυχία, μπορούσε να είναι πιο αδύναμο το ευρώ. Ε, ποια είναι τα εμπόδια για ένα πιο αδύναμο ευρώ και τι μπορείτε να κάνετε για να πετύχετε το στόχο του πληθωρισμού του 2%. Ευχαριστώ. λέει ο Ντράγκη. Η ισοτιμία δεν είναι στόχος μας, στόχος της πολιτικής μας, αλλά η σταθερότητα των τιμών. Αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε εντολή. Όμως η ισοτιμία είναι σημαντική Πρώτα απ' όλα για τη σταθερότητα των τιμών, διότι όταν αναφέρουμε σταθερότητα τιμών, είναι αμφίδρομη η σχέση. Όποτε απέχουμε από το 2% ή κοντά αλλά κάτω το 2%, ε, θέτουμε το πρόβλημα να πετύχουμε τη σταθερότητα των τιμών. Για τη σταθερότητα τιμών και την ανάπτυξη είναι σημαντικό στοιχείο. Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησής μας είναι η ισοτιμία, όταν αποφασίζουμε την νομισματική πολιτική όσον αφορά τις προβλέψεις ε, μεσοπρόθεσμα για τις τιμές, τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τις τιμές. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω φιλανδικά. Υπάρχουν κάποια εμπόδια ούτως ώστε να θέσετε το στόχο του 2% του πληθωρισμού, να το πετύχετε σε ταχύτερο, με ταχύτερου ρυθμού, δηλαδή να τεθεί το 2% σαν ποσοστό πληθωρισμού, σαν μεσοπρόθεσμο στόχο. Απάντηση. Ε, η νομισματική μα πολιτική είναι πολύ ελαστική ε, και υπήρξε επί μακρόν. Στην αρχική μου παρέμβαση είπα ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια Εφαρμόσαμε πολλές δράσεις όσον αφορά την νομισματική πολιτική προς παρόμοια κατεύθυνση. Η νομισματική πολιτική να είναι πιο ελαστική και να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές ε, εξελίξεις. Ο πληθωρισμός είναι κάτω από το 2% και εξήγησα γιατί. Και γιατί θεωρούμε ότι μεσοπρόθεσμα θα συγκλίνει προς τις προσδοκίες προς τις προβλέψεις που είναι σταθερές μέσω μακροπρόθεσμα οι προβλέψεις και ο στόχος μας είναι 2%. Για το ΕΛΚ, ο Πάμπλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αν ήταν 3% πληθωρισμό σήμερα, είχαμε ανάπτυξη, πιστώσεις, κανένα πρόβλημα, είμαι σίγουρος ότι θα σας επικροτούσε το σώμα εδώ. Όμως σήμερα η κατάσταση δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Γιατί έχουμε έναν πληθωρισμό ενάμιση μέχρι το 2018 σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο. Οπότε οι ερωτήσεις μου είναι Συμφωνείτε με αυτή την πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αν ναι, πιστεύετε ότι έτσι εσείς φερέτε σε πέρα στην αποστολή σας. Δεύτερον, τι επιπλέον ε, συστατικά θετικά ή τέλος πάντων μη αρνητικά θα έπρεπε να υπάρχουν στην οικονομία μας ώστε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είσαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να δράσετε. Και τρίτον, ξανά η δεύτερη ερώτηση. Λέω, τι αρνητικό ή τέλο πάντων μη θετικό στοιχείο οικονομικά μιλώντας θα έπρεπε να έχουμε πέρα δηλαδή από τη μίση των πιστώσεων, το χαμηλό ε, πληθωρισμό και την χαμηλή ανάπτυξη στην ύφεση. Τι άλλο θέλετε δηλαδή ώστε να είσαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να πάρετε μη συμβατικά μέτρα ώστε να πετυχαίνετε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τρίτον, Σας ρωτήσαν και άλλοι για την αγορά ομολόγων. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι παραπάνω? Ευχαριστώ. Απάντηση. Δυστυχώς, οι ερωτήσεις σας έρχονται στα πλαίσια της απαγόρευσης που έχω να συζητήσω για την νομισματική πολιτική σήμερα. Αλλά όλα τα εργαλεία, ακόμα και αυτά τα οποία εσείς αναφέρατε, επειδή είμαστε σε προκλογική περίοδο, στην ε, πραγματικότητα πρέπει τα εργαλεία αυτά να τα δούμε σαν ε, απάντηση στις συγκυρίες. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι τα εργαλεία από μόνα τους δεν είναι τέλεια και χρησιμοποιούμε το ένα με το άλλο. Η χρήση τους ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες συγκυρίες σε μια συγκεκριμένη οικονομική και νομισματική κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο και να σχολιάσω περισσότερο γιατί Καταλαβαίνετε ότι αυτό αντιφάσκει με τις αποφάσεις που θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη. Και όσον αφορά τις προβλέψεις του Διεθνούς Μεσοτικού Τεμίου για τον πληθωρισμό που λέει ότι μέχρι το 2018 θα μείνει στο 1,5%, συμφωνείτε? Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα δημοσιεύσει τις προβλέψεις του, τα προγνωστικά του δηλαδή ακριβώς την Τετάρτη στην συνάντηση, ή μάλλον Πέμπτη, Πέμπτη θα ανακοινωθούν. Και θα είναι η πρώτη φορά που το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα δημοσιεύσει προγνωστικά μέχρι το 2016. Οπότε τότε θα απαντηθεί η ερώτησή σας, την Πέμπτη. Λοιπόν, υπομονή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ωραία, εσεί μπορεί να δυσκολεύεστε, εμεί δεν δυσκολευόμαστε όμω και γι' αυτό σα πιέζουμε όσο μπορούμε για να μα απαντήσετε. Μάρκος Φέρμπερ, από το ΕΛΚ τώρα. Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Α, βαβαρικά, ναι, για σένα. Όπως το προηγούμενο Σάββατο στο ποδόσφαιρο σχόλιο προς κάποιον άλλο. Έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αντίθετα με αυτά που είπε ο κύριος Επίνκ. Α, δεν κέρδισε τον όγρο. Δηλαδή τα επιτόκια για τα κρατικά δάνεια έχουν μειωθεί και πάλι για, τη, για την Νότια Ευρώπη δηλαδή σε επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση. Εν προκειμένου ερώτηση. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον ισολογισμό της, δηλαδή θα βγάλει από το χαρτοφυλάκιό της και άλλα χαρτιά. Είχε φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορείτε να πείτε ότι μπορείτε να μείνετε εκεί. Και δεύτερο, ως εποπτεία των τραπεζών εσείς προετοιμάζετε τώρα τις δοκιμές αντοχής και εν πάση περιπτώσει εντατικά. Ακούω δε ότι ορισμένες τράπεζες θα κριθούν σύμφωνα με τους ισολογισμούς τους και άλλες σύμφωνα με τις προοπτικές ισολογισμών. Ερωτώ εγώ, είναι δυνατόν να προκύψει κάποιο λογικό αποτέλεσμα όταν άλλες τράπεζες θα κριθούν στη βάση κλεισμένων ισολογισμών και άλλες ε, στη βάση προοπτικών για τους ισολογισμούς στο μέλλον. ο πρόεδρος Ντάγκη. Για τη δεύτερη ερώτησή σας πρώτα, όλες οι τράπεζες θα κρυφθούν με τον ίδιο τρόπο. Θα γίνει δηλαδή asset quality review, επανεξέταση δηλαδή των στοιχείων του ενεργητικού τους και της ποιότητάς τους, δηλαδή της ποιότητας των ισολογισμών όλων των τραπεζών με τον ίδιο τρόπο, όχι ορισμένες για προοπτικές και άλλες κλεισμένους ισολογισμούς και έχω, το έχω πει από την αρχή ότι αυτή η επανεξέταση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού έχει κάποιο νόημα μόνο εφόσον είναι διαφανής και αυστηρή διότι ο σκοπός εδώ είναι να δοθεί μια αξιόπιστη εικόνα των ισολογισμών του τραπεζικού μας συστήματος στην Ευρωζώνη. ώστε ο ιδιωτικός τομέας να θεωρήσει ότι είναι σκόπιμο να επενδύσει, διότι διστάζει τώρα να επενδύσει σε πράγματα που γι' αυτό είναι άγνωστα και γι' αυτό η asset quality review είναι τόσο σημαντική. Είναι όμως σημαντική και θα είναι αποτελεσματική μοναχά εφόσον είναι διαφανής και μοναχά εφόσον είναι και συνεπής σε όλο το φάσμα τραπεζών της ζώνης ευρώ. Όταν λέω όλες τις τράπεζες ενώ όλες εκείνες που υπάγονται στην άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως και οι μικρές τράπεζες υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς εποπτείας. Η διαφορά μεταξύ της εποπτείας των μεγάλων τραπεζών και των μικρών τραπεζών είναι η ένταση, η εντατικότητα με την οποία οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα εμπλέκονται στην εποπτεία. Για τις 128-130 μεγαλύτερες τράπεζες θα είναι το κέντρο και με τη βοήθεια των εθνικών αρμοδιών αρχών και ανεξαρτήτων μερών και των μικτών ομάδων επιθεωρητών που θα ε, προέρχονται από διαφορετικές δικαιοδοσίες εποπτείας από διάφορες, ε, από διάφορες χώρες της Ένωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός διαφάνειας. Για τις μικρότερες τράπεζες βέβαια το εθνικό στοιχείο της εθνικής αρχής θα είναι μεγαλύτερο αναλογικά όμως το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, επιφυλάσσει σε αυτό το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία και ενδεχομένως να επεμβαίνει και το ίδιο. Άρα ίση όρια ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Για την πρώτη σα ερώτηση, σα παρακαλώ την επαναλάβετε, γιατί δεν την κατενόησα απολύτω. Η κεντρική τράπεζα είναι διατεθειμένη να φέρει ξανά στις αγορές κρατικά ομόλογα, αφού τώρα το επίπεδο των επιτοκίων στη ζώνη ευρώ έχει κατέλθει και μάλιστα σημαντικά. ο Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι μια πραγματική, η SMP Holdings, ομόλογα που έχουν αγοραστεί όταν άρχισε το Securities Markets Program. Και η δέσμευση που είχε αναλυφθεί τότε, δηλαδή το 2010 αν θυμούμε καλά, ήταν να κρατηθούν τα ομόλογα αυτά μέχρι την ορίμανσή τους. Στο μεταξύ τα ομόλογα αυτά έχουν πέσει διότι έχουν περάσει την ορίμανση και το ίδιο το πρόγραμμα λοιπόν έχει μειωθεί γιατί όταν φτάνουν στην ορίμανση δεν αντικαθίστανται δηλαδή. Η άλλη περίπτωση είναι η θεωρητική που δεν επήλθε ποτέ δηλαδή για τα ομόλογα που αγοράστηκαν υπό την ισχύ του OMT. Οπότε αυτά αγοράζονται και πολλούνται, άρα εκεί δεν υπάρχει καμιά δέσμευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές Βαν Κοκ. Ευχαριστώ Σάρων. Κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσεις μου θα αφορούν τις δράσεις της Τρόικας. Συνοψίσατε σε αυτά που είπατε τη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την τελευταία πέντα ετία και όπως είπατε όταν το πρόγραμμα αποφασίστηκε το OMT, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατάφερε να αντιμετωπίσει τις κερδοσκοπικές πιέσεις όσον αφορά τα κρατικά, το κρατικό χρέος. Νομίζετε ότι αν το πρόγραμμα OMT είχε ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είχε αποφύγει το να επηρεάσει η ελληνική κρίση την Κύπρο και την ε, ε, Πορτογαλία παραδείγματος χάρη. Είπατε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη τώρα από ότι το 2009. Βλέποντας όμως τα μακροοικονομικά στοιχεία ανησυχούμε. Διότι το ποσοστό κατοικού χρέους όσον αφορά το ΑΕΠ είναι πάνω από το 120% και το Εθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι πάνω από 120% δεν είναι βιώσιμο ποσοστό και κυρίως στην περίπτωση της Ελλάδος ε, η κυρία Λαγκάρτ προτείνει μέτρα τώρα στον αφορά το χρέος του ελληνικό. Αν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα και να αποφασιστούν κάποια μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δεχτεί απώλειες διότι στην πρώτη αναδιάθρωση του χρέους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ανέλαβε τις απώλειες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα έχει 34 δισεκατομμύρια του ελληνικού κρατικού χρέους. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει αυτές τις απώλειες, μπορεί, μπορούν να αποφευθούν προβλήματα οι Έλληνες πολίτες στις ελληνικές τράπεζες. Και αυτό θα ήταν χρήσιμο σήμερα όταν δεν υπάρχει πίεση από τον πληθωρισμό και δεν υπάρχουν κάποιες προσδοκίες για αύξηση του πληθωρισμού. Ε, ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό. Να απαντήσω πρώτα στην πρώτη ερώτηση. Η γενική απάντηση είναι ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα. Και αυτό πάντα αληθεύει εκ των υστέρων. Όμως υπάρχει και μία πιο βαθιά απάντηση. Αν διερωτηθούμε, ποιοι παράγοντες επανέφεραν την αξιοπιστία στο ευρώ, δημιούργησαν εμπιστοσύνη από πλευρά του υπολείπου κόσμου προς το ευρώ. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε επί τριών στοιχείων. Πρώτον, το πώς πολλές χώρες, κυρίως αυτές που υπέστησαν τα προβλήματα, πώς ε, έλαβαν μέτρα για βελτίωση των οικονομικών τους πολιτικών και έγιναν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες αναμόρφωσης μεταρρύθμισης. Σε πολλές χώρες έγινε προσπάθειες πριν από τον Ιούλιο του 2012. Και σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίστηκαν οι προσπάθειες και μετά. Αυτός ήταν ένας παράγοντας, ο δεύτερος παράγοντας, που συχνά τον λησμονούμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012, το οποίο ξεκίνησε τις προσπάθειες για Τραπεζική Ένωση. Τρίτο στοιχείο η εκκίνηση του προγράμματος OMT. Αυτοί οι τρεις παράγοντες διαπλέκονται και παίζουν ένα σημαντικότατο και αποτελεσματικότατο ρόλο. Συνέτειναν στο να υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη προς το ευρώ. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο ερώτημα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, είπα. Δεν είπα ότι είναι καλή, είπα είναι καλύτερη. Καλύτερη από ό,τι κατά το παρελθόν. Σίγουρα όμως δεν είναι καλή. Η ανεργία είναι πολύ ψηλή. Όσον αφορά την ανεργία, είχαμε κάποια πολύ μικρά σημάδια βελτίωσης. Σταθεροποιείται τους τελευταίους μήνες και σε κάποιες χώρες με προβλήματα μειώνεται. Η Πορτογαλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Μειώθηκε κατά 2% η ανεργία και σταμάτησε η μείωση της απασχόλησης. Έχουμε κάποια σημάδια. Αλλά θα πρέπει εδώ να θέσουμε το εξής ερώτημα. Γιατί αυξήθηκε η ανεργία τόσο πολύ σε κάποιες χώρες και πολύ λιγότερο σε άλλες. Έχουμε μία υποψία ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό διαθροτικής ανεργίας μέσα στο 12% της ανεργίας για να δούμε μια σημαντική, πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας, όχι μόνο η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά χρειάζονται σοβαρές με διαθροτικές μεταρρυθμίσεις σε αρκετά κράτη-μέλη της ε, Ευρωζώνης. Τέλος, κατά πώς επομίζεται τις απώλειες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή όχι Τώρα για την ανακούφιση του χρέους ε, δεν πρέπει να κάνουμε εικασίες τώρα, αλλά να πούμε κάτι που ισχύει. Δεν μπορούμε να προβούμε σε νομισματική χρηματοδότηση. Το άρθρο 123 απαγορεύει τη χρηματοδότηση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε εικασίες όσον αφορά τη διευκόλυνση του χρέους. Όσον αφορά την Ελλάδα και άλλες χώρες, ειδικά για την Ελλάδα, Πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε επί της εφαρμογής, πλήρους εφαρμογής του προγράμματος. Καλώς. Η άμεση διαχείριση και η κατά βέβαια έχει διαφορά. Εκ μέρους του ΕΛΚ τώρα, και η Μίτσελ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ Πρόεδρε Ντράγκη Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις παρακαλώ. Η πρώτη έχει να κάνει με τον τραπεζικό δανεισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρατε ότι στο πλουστάσιό σας, στον κατάλογό σας, δεν ξέρω τι από τα δύο είπατε τελικά, έχετε διάφορα εργαλεία. Θα ήθελα όμως συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να οδηγηθούν σε έναν αυτοματισμό δανειοδότησης που δεν τον έχουν σήμερα. Διότι είναι δημόσιο χρηματοπιστωτικά μάλλον ιδρύματα τα οποία όμως δεν δρούν έτσι αυτόματα δημοσιονομικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτοματισμό, τουλάχιστον στη δικιά μου τη χώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πια παραδοσιακή τραπεζική διαχείριση μπορεί δύο ίδιες ηλικίες άνθρωποι με την ίδια διοκτησία, ίδια εισοδήματα να πάνε σε δύο τράπεζες και ένας μπορεί να περάσει ώρες και άλλος μπορεί πολύ πιο γρήγορα να προχωρήσει αυτά που θέλει. Μπορούμε λοιπόν παρακαλώ να ε, βρούμε πάλι αυτούς οι οποίοι παίρνουν ε, τις αποφάσεις στις τράπεζες για τη διανυδότηση και να τους βάλουμε να ανταποκρίνονται σε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και να δρουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων. Δεύτερον, Ρωτούσα τον προκάτοχό σας όσον αφορά τον πληθωρισμό σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, με το ενεργητικό. Στο Δουβλίνο τουλάχιστον έχουμε τεράστιο πληθωρισμό ε, στις κατοικίες. Τι θα γίνει με αυτό. Δράγκη. Θα αρχίσω από τη δεύτερη ερώτησή σας. Υπάρχουν δείγματα αύξησης τιμών κατοικιών σε κάποια μέρη της Ευρωζώνης. Τα παρατηρούμε με προσοχή τα φαινόμενα αυτά. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι την προηγούμενη φορά. Πρώτα απ' όλα ότι οι πιστώσεις είναι πολύ χαμηλές. Και όταν είχαμε μεγάλη αύξηση στον τιμό την προηγούμενη φορά, τότε οι πιστώσεις, αν μη τι άλλο, έρεαν άφθονα. Συνεπώς, ναι, πολύ νωρίς να μιλήσουμε για φούσκα στο στεγαστικό τομέα. Πάντως, παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση σίγουρα δεν είναι να αλλάξουμε την νομισματική μας πολιτική, γιατί η νομισματική μας πολιτική έχει να κάνει με τη σταθερότητα τιμών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Η απάντηση είναι να έχουμε ένα μέσο στη διάθεσή μας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τοπικές φούσκες. Και οι τοπικές φούσκες αντιμετωπίζονται με τοπικά εργαλεία, δηλαδή μικροεποπτικά. Γι' αυτό η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός τέτοιων υποπτικών εργαλείων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι αυτό που βοηθάει στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Και παγώνει την νομισματική πολιτική και την αναγκάζει να μην ε, κυνηγάει στόχους που δεν εμπίπτουν στην εντολή της. Η άλλη σας ερώτηση τώρα έχει με τη συμπεριφορά των τραπεζιτών και των τραπεζών. Έχετε δίκιο. Ο δανεισμός, όπως λέει και ο κλάδος, έχει γίνει κάτι σαν ε, αυτόματος πιλότος αντί να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει όπως θα έκανε κάποιος τραπεζίτης πριν από όχι πάρα πολλά ε, χρόνια και να δει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό βέβαια κοστίζει στον τραπεζικό τομέα και σημαίνει ότι η ανάλυση για τις πιστώσεις δεν γίνεται τόσο ανάλογα με αυτόν που έχουν απέναντί τους, αλλά είναι κάτι γενικό. Το αποτέλεσμα μερικές φορές είναι να δώσουν σε κάποιον πιστώσει σε κάποιον που δεν θα έπρεπε να δώσουν και να μην δώσουν σε κάποιον που θα έπρεπε να δώσουν. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και πλήτη και την κερδοσκοπία της τράπεζας, αλλά είναι και πολύ πιο σοβαρό μερικές φορές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τον, για λόγο με το, που εξηγεί μάλλον τη συμπεριφορά αυτή των τραπεζών. Οι περισσότεροι τραπεζίτέ το καταλαβαίνουν σήμερα. Ήταν μια εξέλιξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2010, αυτή τη δεκαετία. Άλλαξε η συμπεριφορά των τραπεζών. Σκέφτονται αλλιώ σήμερα. φταίνει οι συνθήκες που επικρατούσαν πριν την κρίση σε έναν βαθμό. Ενώ σήμερα η εντύπωση που έχει κανείς είναι ότι σκέφτονται πολύ περισσότερο για το πώς θα δίνουν πιστώσεις, όχι έτσι γενικά και χωρίς κριτήρια. Η διαδικασία είναι από τη φύση της τέτοια που κάνει τις τράπεζες ε, να δίνουν δάνεια χωρίς να σκέφτονται συγκεκριμένες παραμέτρους και κριτήρια. Τα ενυπόθηκα δάνεια, ας πούμε, ήταν κάτι έτσι γενικό. Οι πιστώσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλου είδους δάνεια δεν μπορεί να δίνονται με αυτόματο πιλότο. Ευχαριστώ. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τόσο ενδιαφέρουσε ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Λεωνάρντο Ντομένιτσι από τους σοσιαλιστές. Πρόεδρε, για την τελευταία σας αυτή εμφάνιση κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας θα σας θέσω μια ερώτηση γενική. Πιστεύω βλέπετε ότι κά... με κάποια έννοια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεπέρασε τις αρμοδιότητές της. Αλλά δεν είναι πρόκληση αυτό δεν παρεύει τις συνθήκες και δεν νομίζω ότι είσαστε εσείς ο James Bond. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε και τη δουλειά άλλων. Διότι από όλους τους θεσμούς, αυτός ο θεσμός υπερασπίστηκε με βασιστικότητα την εκαιρεότητα της Ευρωζώνης και κράτησε στη ζωή ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης που κινδύνευε να κατακαιρματιστεί. Πολύ συχνά εσείς και άλλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπατε ότι οι τεχνικοί, οι τεχνοκράτες έχουν τα ωριά τους, πρέπει να παρέμβει πολιτική. Ερώτηση, τι είδου μήνυμα δίνει ο πολίτης, Ευρωπαίος πολίτης Μάριο Ντράγκη που πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο μήνυμα θα ήθελε να βγει τώρα στην προκλητική εκστρατεία. Δεν μιλάω για προγράμματα, για πώληση, για αρχιτεκτονικέ θεσμών και μεταρρυθμίσει διαθροτικέ σε εθνικό επίπεδο. Μιλώ για κοινή νοοτροπία, νοοτροπία. Ε, Πώ να ξαναπροωθήσουμε και να δώσουμε ορμή σε ένα πρόγραμμα που οδηγεί σε more perfect union, σε μια πιο τέλεια πολιτική ένωση στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Απάντηση. Δεν είναι απλή ερώτηση για έναν ταπεινό εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας, για έναν τραπεζίτη και έναν γραφειοκράτη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση υπό μια ασθενή νοτροπία, τη δική μου νοτροπία. Τι πρέπει να κάνει η Ένωση, πού πρέπει να επανέλθουν. Πρέπει να επανέλθουμε η Ένωση να ξαναγίνει μια ε, νήσος ευημερία, ένα νησί ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ένα μέρος ανάπτυξης στον κόσμο, ένας τόπος στον κόσμο όπου ε, απολαμβάνει κανείς να είναι. Έχει γούστο να βρίσκεται κανείς εκεί, όπου υπάρχουν ελπίδες, και για να γίνει αυτό δεν θα ήθελα να μαντέψω ποιου είδους πολιτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν διότι δεν μπορώ να πω κάτι ενδιαφέρον πάνω σε αυτό. Υπάρχουν τομείς όπως οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, η σταθερότητα στα πολιτικά συστήματα, όπως κοινή βούληση για ανάπτυξη, όχι για να ξεφύγουμε από το χρέος, διότι αν ανακαλύψαμε κάτι, αν κάποιο μάθημα βγήκε και που έμαθε η Ευρώπη και η Ευρωζώνη, είναι το εξής, ότι το, μια τέρμονη δημιουργία χρέους δεν δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη. Σε κάποια φάση επέρχεται ύφεση. Και όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια η ύφεση είναι πάρα πολύ οδυνηρή. Όχι μόνο λόγω των αμέσων αποτελεσμάτων αλλά και επειδή γκρεμίζονται ελπίδες κυρίως για τους νέους. Αυτό θα έλεγα. Το μήνυμα είναι της ανοικοδόμησης. Ανοικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να γίνει ένα νησί ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ελπίδων, ελευθερίας. Ευχαριστώ. Καλώς λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άστριντ. Η Άστριντ Λούλινγκ για το ΕΛ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη. Είχα σημαντική συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ήθελα να σας θέσω τρεις ερωτήσεις κύριε Ντράγκη. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο για να μελετήσω την Πολιτική Ένωση, για να σπουδάσω, έμαθα ότι χαμηλός πληθωρισμός ήταν κάτι καλό. Πράγματι ε, πέρασαν ήδη σχεδόν 60 χρόνια από τότε. Δεν είναι δυνατόν λέει ο κύριος Ντράγκη. Σίγουρα με έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Αλλά πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής διότι στη χώρα μου το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου ο πληθωρισμός επιτέλους είναι κάτω από το 2% λόγω της ε, προσαρμογής μας, της τιμαριθμικής προσαρμογής μας και πιστεύω ότι αυτό θα, θα ήταν καλό αν το 2014 ε, μπορούμε να καλύψουμε το 2,5% να καλύψουμε τους ελάχιστους μισθούς συντάξεις και λοιπά, δημόσιου τομέα. Αν πετύχουμε το 2,5% στους μισθούς και λοιπά. Ήτανε ο προκάτοχός σας, ο κύριος Τρισέ, πάντα επέμενε λέγοντας μας ότι πρέπει να καταργήσουμε την αυτόματη τη αριθμική α, μετα, αλλαγή, μεταβολή, αναπροσαρμογή. δεν θα πρέπει να μιλάμε για τον αποπληθωρισμό. Λοιπόν, άρα πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό. Η ισοτιμία του κινέζικου νομίσματος αυξήθηκε σε σχέση με το ευρώ και το δολάριο. Νομίζω ότι τελευταία χρόνια αυξήθηκε πάνω από 25%. Τις τελευταίες μέρες όμως μειώθηκε η ισοτιμία για ποιο λόγο μπορείτε να το εξηγήσετε. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί, ότι είναι σκόπιμο από πλευράς των κινέζικων αρχών επιδιώκεται αυτός ο στόχος. Μετά από την ε, γνωμική νομοδότηση του Συμβουλίου όσον αφορά τον φόρο των χρηματοστικών συναλλαγών δεν πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της σχετικά με τη θέσπιση αυτού του μέτρου στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας που θα έπληκτε πολλές υπηρεσίες της Ευρώπης. Είπατε λοιπόν εσείς ότι ο στόχος ήταν μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνέπειες αυτού του φόρου θα ήταν αντίθετες. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεχώς με την υποβολή ερωτήσεων και μάλλον και την, ε, τις θα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε στο δίλεπτο. Ευχαριστώ λέει ο κ. Δράκη. Τι είναι αυτό? Α, όταν λέμε ότι αυτό που οθεί την ανάκαμψη τώρα ποιο είναι. Παλιά κυρίως από τις εξαγωγές οδηγεί το κατ' παρελθόν. Τώρα σταδιακά ε, προωθείται η ανάκαμψη και από την εσωτερική ζήτηση. Άλλες κινητήρες δυνάμεις είναι η νομισματική πολιτική και η αποκατάσταση εμπιστοσύνη. Αλλά, και εκεί συμφωνώ μαζί σας, άλλος κινητήρας για την ανάκαμψη είναι ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών, των ημερομισθείων και των συντάξεων, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ένα το ποσοστό των συνταξιούχων στην Ευρωζώνη είναι αρκετά υψηλό. Λοιπόν, η αγοραστική δύναμη διατηρείται υψηλή λόγω χαμηλού πληθωρισμού. Από αυτή την έποψη πρέπει να το δούμε. Έχουμε χαμηλή τιμή ενέργειας και τροφίμων. Ε, τουλάχιστον πληθωρισμό αυτά. Ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος από ότι κατά το παρελθόν είναι κάτι που υποστηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη πλευρά έχουμε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Άρα το πραγματικό εισόδημα των νέων του και των ανέργων είναι ε, χαμηλή η αγοραστική τους δύναμη. Άρα δεν μπορεί να στηρίξει αγοραστική αυτή δύναμη την ανάκαμψη. Η δεύτερη ερώτηση. Δεν έχω ιδέα, πρέπει να κοιτάξω τι είπατε, γιατί, γιατί πρώτα αυξήθηκε το ποσοστό και μετά μειώθηκε. Για το κινέζικο νόμισμα δεν ξέρω γιατί αυξήθηκε η ισοτιμία του και μετά μειώθηκε. Είναι πολύ περίπλοκη η κινέζικη οικονομία. Δεν ξέρω την απάντηση. Όσον αφορά το φόρο ε, συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θέλει να σχολιάσει διότι αυτό εμπίπτει 100% εντός των αρμοδιοτήτων των κυβερνήσεων και των πολιτικών αρχών. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πτυχές του φόρου αυτού που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη διαμόρφωση νομισματικής μας πολιτικής και εμείς συνεργαζόμασταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να διορθώσουμε αυτές τις αρνητικές πτυχές της ε, πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα οι σοσιαλιστές. Άντωνη Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για όλα όσα κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Πήρατε σημαντικές πρωτοβουλίες και πετύχατε σήμερα η Ευρώπη να μην βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Αλλά όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, οι πολίτες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουν από αυτήν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Δυστυχώ, είμαστε πολύ μακριά από αυτό ακόμα. Σήμερα υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο για την νομισματική πολιτική. Εξού και ερωτήσει μου. Πρώτα απ' όλα για την νομισματική πολιτική. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ε, περισσότερα περιθώρια στα πλαίσια της νομισματικής αυτής πολιτικής. Και δεύτερον, πώς πετυχαίνει η νομισματική μας πολιτική του στόχου της Ένωσης. Από την ΦΕΔ ακούσαμε πρόσφατα για την ε, αϊφόρο απασχόληση και πώς θα είναι συμβατή με την νομισματική πολιτική. Λοιπόν, εδώ στην Ευρώπη πώς εφαρμόζεται αυτό. Δηλαδή η δικιά μας νομισματική πολιτική συνάδει με τους στόχους μας, απασχόληση για παράδειγμα. απάντηση. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη νομισματική πολιτική αυτή τη στιγμή και τις αποφάσεις τις σχετικές δηλαδή, αλλά θα απαντήσω στις άλλες πτυχές των ερωτήσεών σας. Η νομισματική πολιτική έχει κάνει πολλά τα τελευταία δυόμιση χρόνια και εξακολουθεί να βοηθάει. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κάνει είναι τη δουλειά που κανονικά πρέπει να κάνουν άλλοι. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κυβερνήσεις, για παράδειγμα. Και τώρα που έχουμε βγει από τη φάση εκείνης της κρίσης που επιγόντως έπρεπε κάτι να κάνουμε. Τώρα λοιπόν αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι να σκεφτούν και πάλι τις δημοσιονομικές τους προσπάθειες και όχι υπό την έννοια, το λέω αυτό αμέσως σε σχέση με την πρόοδο που έχουν κάνει και τις προσπάθειές τους που βέβαια ήταν τόσο τεράστιες αλλά με την έννοια του να συνεχίσουν αυτό που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ονομάζει φιλική προσπάθεια για απαγίωση της ανάπτυξης. Χαμηλότερη φορολόγηση, μείωση τρέχουσων δαπανών, ε, δεχομένως αύξηση των ε, κατακεφαλήν δαπανών στις υποδομές μεταξύ άλλων. Να ξέρετε ότι οι χώρες ε, και δεν ξέρω πόσα πολλά χρόνια, δέκα χρόνια, είχαν πολύ χαμηλές επενδύσεις στις ε, υποδομές. Τώρα κάθε χώρα πρέπει να δει πού θα δαπανεί στις υποδομές, στις υπηρεσίες, γιατί είναι βασικό κομμάτι αυτής της σταθεροποίησης που θέλουμε. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και ονομάζονται έτσι ακριβώς γιατί εξαρτάται από το σε ποια χώρα αναφερόμαστε. Όλες οι χώρες πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Άλντε, ο Νίλς Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προεβδομάδος η Επιτροπή μας ψήφισε την έκθεση για την Τρόικα με οδηγό την Κομισιόν, συνοδηγό την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το Παγκόσμιο ε, Ταμείο και από πίσω να κάθεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που να οδηγεί το ποδήλατο. Πέστε μας τα σχόλιά σας χωρίς ε, να μας πείτε για το Goldfinger. Τώρα, ο δείχτης Wix του Σικάγο σημαίνει μειωμένη ρευστότητα και επομένως αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα. Αχ, τι ωραία που είπατε για στον Μάρτιν, γιατί ταιριάζει και με τον James Bond. Μην αρχίσουμε πάλι, μην αρχίσουμε πάλι με... Μην το παρακάνουμε με την παραβολή με τον James Bond. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ. Λέει ο πρόεδρος Δράκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχετε δίκιο ότι κάθεται στο πίσω κάθισμα της Τρόικα. Είναι συγκεκριμένη η συμβολή που μπορεί να κάνει στον ε, χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα και όλο και περισσότερο θα γίνεται αυτό στο μέλλον. Υπάρχει λόγος που κάθεται στο κάθισμα η Κεντρική Τράπεζα. Εάν ο διάβλος δανεισμού τραπεζών, που είναι και ο βασικός που έχουμε, δεν λειτουργήσει, τότε η νομισματική μας πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι αποτελεσματική. Άρα η παρουσία, ένα, μάλλον ένας από τους λόγους για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκεί είναι να βελτιώσει τη λειτουργία του διάβλου δανεισμού των τραπεζών ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η νομισματική πολιτική. Συχνά αυτή η βελτίωση δεν περιορίζεται μοναχά στον τραπεζικό τομέα, όμως απαιτεί ενέργειες και σε άλλους τομείς. Όμως αυτή είναι η σκοπιά που υπαγορεύει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα. Για το μέλλον θα δούμε. Ασφαλώς θα ήταν πρόημο να προβληματιστεί κανείς για άλλους ρόλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι να μπορέσουμε να πούμε ότι έχει περάσει η κρίση με κάποιο πιστικό τρόπο. Για το άλλο που είπατε για τη ρευστότητα. Εκεί παρακολουθούμε την κατάσταση της ρευστότητας. Η υπερβάλλουσα ρευστότητα κινείται ή προκαλείται από ένα πλήθος παραγόντων. Και νομίζω δεν είναι εύκολο να καθιερωθεί μια σχέση μεταξύ της υπερβάλλουσας ρευστότητα και της λειτουργίας των αγορών. Εξετάζουμε την υπερβάλλουσα ε, ρευστότητα, την πλεονάζουσα ρευστότητα στα τέλη του μηνός που μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ε, περασμένο VIX. η πρόεδρος Σάρων Ο τελευταίος ομιλητής τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες Πέτερ Σίμον. Κύριε Ντράγκη, να σας ρωτήσω κάτι για άλλο θέμα, για τις προτάσεις σας για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Ο Ευρωπαϊκός Λογαριασμός δηλαδή να συλλέγονται, να προσκαλούνται χρήματα, να συλλέγονται χρήματα με ένα σταθερό επιτόκιο που να το καθορίζει η Κομισιόν ή κάποιος άλλος οργανισμός και με αυτά τα επιτόκια να δίνονται πιστώσεις στις ε, βιομηχανίες. Εγώ, όπως στην Ιταλία η Φεντακάς, τα μικρά ταμιευτήρια που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα βλέπετε στον προβληματισμό της Κομισιόν τον κίνδυνο ενδεχομένως ότι σε αγορές που ζουν από τις business με τις αποταμιεύσεις και το κάνουν αυτό τα ταμιευτήρια. Μήπως εκεί ακριβώς αυτή, αυτός, μήπως δηλαδή υπονομευτεί αυτός ο καταρχήν υγιής μηχανισμός και η οικονομία τελικά όχι μόνο να προωθηθεί λιγότερο ακριβώς διότι αυτοί οι θεσμοί θα χάσουν την βάση τους, θα χάσουν δηλαδή την ικανότητα να δίδουν πιστώσεις. Δεν βλέπετε επίσης τον κίνδυνο σε αγορές όπου οι τράπεζες δεν λειτουργούν καλά να μπουν σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα επειδή θα μειωθούν τα αποθεματικά τους. ο Δεν είμαι και βέβαιος ότι τα μακροπρόθεσμα πιστοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχουν τέτοιο μέγεθος που να προκαλέσουν αυτές τις τεράστιες επιπτώσεις που περιγράφεται στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Το βλέπω σαν ένα από τα μέτρα για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Αλλά δύσκολα το βλέπω σαν κάτι που μπορεί να ανταγωνιστεί με άλλες πηγές χρηματοδότησης του τραπεζικού κλάδου γενικότερα. Από την άποψη αυτή λοιπόν δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λόγος φόβου. Και ε, στον βαθμό που θα υπάρχουν κάποιες περιθωριακές βελτιώσεις της οικονομίας από τις ε, προσπάθειες αυτής της Κομισιόν θα οδηγήσουν και σε μια αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες που προαναφέρατε. Ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώσαμε τον διάλογο για τα νομισματικά θέματα για την ώρα. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ακρόση, αλλά θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Μην φύγετε παρακαλώ. Έχουμε ένα-δύο σημεία να συζητήσουμε και θα επανέλθουμε μετά για την δεύτερη ακρόαση μας. Okay. Okay, let's, let's recommence. Καλώς, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Και περνάμε στην δημόσια ακρόαση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά υπό τον ρόλο του, του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε παρακαλώ τις ερωτήσεις. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν επικαλύψεις και δεν έχουμε και τόσους πολλούς ε, ερωτώντες, οπότε προτείνω να ακολουθήσουμε τη διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή να ακούσουμε την παρουσίαση πρώτα βέβαια του κύριου Ντράγκη, μετά να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά να απαντήσει ο κύριος ε, Ντράγκη συνολικά στις ερωτήσεις αυτές και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά νομίζω ότι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου αυτό είναι προτιμότερο. Λοιπόν, έχετε και πάλι το λόγο κύριε Δράγκη. Ευχαριστώ Σάρον, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ στην συνεδρίαση αυτή για να σας αναφέρω τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του ESRB. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση μετά την δημοσιονομική κρίση μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα δημοσιονομικό πιο εύρωστο. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου σιγά σιγά πετυχαίνει τους στόχους του. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας ενημερώσω για το συνεχιζόμενο έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Από τότε που άρχισε η κρίση έγιναν σημαντικά βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες του δημοσιονομικού συστήματος. Την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς αυτής άρχισαν να ισχύουν νέοι υποπτικοί κανόνες που προσφέρουν ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Και θέλω να αναγνωρίσω εδώ και τον ρόλο κλειδί που έπαιξε το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σημαντικός στόχος. Τώρα με τους νέους εποπτικούς αυτούς κανόνες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να εφαρμόσει μακροεποπτική πολιτική. Προκειμένου να λειτουργεί καλά τώρα βέβαια η πολιτική αυτή, μένουν πολλά να γίνουν από τη δικιά μας την πλευρά, γιατί εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σα ενημερώσω ότι από την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ στην Επιτροπή σα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έκανε σημαντικά βήματα για να ανταποκριθεί στις προκλήσει αυτέ. Τώρα που μιλάμε, ε, δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μα διάφορα έγγραφα που έχουν να κάνουν με το πώ οι διάφορε αρχέ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μακροεποπτικά εργαλεία σύμφωνα με τους νέους εποπτικούς κανόνες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι σχετικά με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και ελπίζουμε οι διάφορες αρχές το υλικό αυτό να το βρούνε χρήσιμο και να τους βοηθήσει στην δικιά τους πολιτική και πολιτικές δράσεις. Βέβαια πρέπει να βγούμε ακόμα περισσότερο από την κρίση. Και η μακροεποπτική πολιτική βοηθάει ακριβώς να έχουμε στη διάθεσή μας την κατάλληλη προστασία. Όμως η χρήση μακροεποπτικών μέσων θα είναι κάτι χρήσιμο και στο εγγύς μέλλον, αλλά και αργότερα. Υπάρχουν αρχές κάποιων χωρών που ανησυχούν πολύ για το θέμα της μόχλευσης και της ε, ανάπτυξης στον ε, τομέα των ε, οικοδομικών των κατοικιών και πολλές χώρες έχουν ήδη ενεργοποιήσει μακροεποπτικά μέσα. Για παράδειγμα η Σουηδία εισήγαγε ένα όριο στάθμισης κινδύνου για υποθήκες και μέτρα μακρορευστότητας. Οι κάτω χώρες από τη δικιά τους την πλευρά ενεργοποίησαν ένα δίχτυ σχέσης δανείου αξίας για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους δυσκολίες στο στεγαστικό τομέα. Συγχρόνως στο Ηνωμένο Βασίλειο η Τράπεζα της Αγγλίας και το θησαυροφυλάκιο της χώρας Επίσης έχει προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα που το λέει Funding for Lending, δηλαδή χρηματοδότηση για δανεισμό. Και μόλις πριν από μερικές εβδομάδες η γερμανική Bundesbank εξέφρασε ανησυχίες για τις εξελίξεις όσον αφορά στην κρίση του στεγαστικού τομέα σε μεγάλες γερμανικές πόλεις. Θέλω τώρα να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες όσον αφορά το υλικό το οποίο δημοσιεύουμε. Και ξεκινάω λέγοντας ότι τα έγγραφα αυτά είναι η τρίτη σημαντική συνεισφορά μας καταλητική για την ανάπτυξη του μακροεποπτικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να θυμόσαστε ότι το 2012 είχαμε μια πρώτη σύσταση προς τα κράτη-μέλη όπου προτείναμε τη δημιουργία εθνικών αρχών με μακροεποπτική εντολή. Συνεχίζουμε βέβαια να αξιολογούμε την κατάσταση, αλλά μπορώ ήδη από τώρα να σας πω ότι η σύσταση αυτή οδήγησε σε ένα κύμα νομοθετικών πρωτοβουλειών στις χώρες μέλη. Σήμερα 19 χώρες μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει μακροεποπτική νομοθεσία, ενώ συγχρόνως υπάρχουν διάφορα νομοσχέδια σε άλλα 7 κοινοβούλια, σε άλλες 7 χώρες. Πέρυσι μάλιστα στηρίξαμε την σύσταση αυτή με μία νέα για να προσφέρουμε στις εθνικές μακροεποπτικές αρχές τα κατάλληλα μέσα να φέρουν σε πέρα στην εντολή τους. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές αυτές έχουν στη διαθεσή τους τα κατάλληλα μέσα για να πετύχουν ενδιάμεσους στόχους που τελικά θα συνεισφέρουν στη δημοσιονομική σταθερότητα. Συμπεριλαμβάνουν στόχους όπως ε, να αποφεύγουμε, να μειώνουμε την ε, υπερβολική αύξηση χρεών, την μόχλευση, τις ε, διάφορες ασυμμετρίες στην ληξιμότητα κλπ. Έτσι προχωράμε περισσότερο στην μακροποπτική μας πολιτική. Ένα βασικό στοιχείο πάντως του υλικού μας είναι ένα εγχειρίδιο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις εθνικές μακροεποπτικές αρχές και δίνει συμβουλές για το πώς να σχεδιάσουμε και πώς να θέσουμε σε εφαρμογή μακροεποπτικές πολιτικές στον τραπεζικό τομέα. Το αρχιερίδιο αυτό συνοδεύεται και από μια μικρή έκθεση, εμβληματική θα λέγαμε, που προσφέρει μια γενικότερη παρουσίαση για την λειτουργία των μακροοικονομικών αυτών εργαλειών. Επίσης, βλέπουμε στην τη βλέπουμε στην έκθεση αυτή σαν ένα εργαλείο που θα βοηθήσει πολύ στην ε, ενημέρωση της μακροεποπτικής πολιτικής, ενημέρωση προς τους πολίτες δηλαδή, σε μια γλώσσα πραγματικά κατανοητή. Και εδώ περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία, είτε το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθυμα ασφάλειας, είτε άλλα εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν με συστημικές τράπεζες και διαρθρωτικούς κινδύνους. Αναφέρουμε συνέχεια τα εργαλεία αυτά ώστε να καλύπτουν τους στόχους για τους οποίους προορίζονται και βλέπουμε πώς χρησιμοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πότε να ενεργοποιηθούν, πότε να απενεργοποιηθούν κτλ. Το εγχειρίδιο επίσης αναφέρεται και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με όλα τα εργαλεία αυτά, τα επιμέρους εργαλεία. Για παράδειγμα, πώς να επιλέξει κανείς το πιο κατάλληλο εργαλείο για ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Πώς να ε, μειώσει την τάση που υπάρχει για δράνεια από τις αρχές κάθε φορά που οι αρχές πρέπει να ξοδέψουν αμέσως, αλλά θα υποφεληθούν από ένα τέτοιο μέσο πολύ αργότερα. Πώς επίσης να μεταφέρουμε στο ευρύ κοινό τα περί μακροποπτικής μας πολιτικής και τέλος πώς να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις σε άλλες χώρες άπαξ και χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Μάλιστα αυτό το τελευταίο με φέρνει τώρα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Έχουμε νέο ρόλο, νέες αρμοδιότητες πέρα από την γενική μας ε, αρμοδιότητα που είναι οι συστάσεις και οι προειδοποίησεις. Οι νέες αυτές αρμοδιότητες είναι κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις για συγκεκριμένα μακροεποπτικά μέσα. Ε, μας ζητάνε επίσης να συμμετέχουμε και στη διαβούλευση όσον αφορά την αναθεώρηση των υποπτικών κανόνων. Πρέπει βέβαια να έχουμε στη διάθεσή μας στέρες, υποδομές και οικονομικό πλαίσιο για να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά και εδώ είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα η οποία θα βοηθήσει με τα διάφορα μέτρα μακροεποπτικής πολιτικής ώστε να υπάρχει ενημέρωση και θα βοηθήσει η ομάδα αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, να ετοιμαστεί καλύτερα. Δουλεύουμε περισσότερο πάνω σε γραμμές προς τις αρχές, προετοιμάζοντας τα στοιχεία για το αντικυκλικό κεφαλαικό απόθεμα ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, θα ολοκληρώσω Κοιτώντα λιγάκι προς το μέλλον, ποιες είναι οι προκλήσεις κλειδί για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Οι επιπλέον αρμοδιότητές μας υπό τους εποπτικούς κανόνες μας υποχρεώνουν να ενισχύσουμε την ανάλυση της πολιτικής μας και του συστημικού κινδύνου. Ενισχύεται επίσης ο εποπτικός μας ρόλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως, πρέπει να εξετάσουμε την διαδικασία λήψεων αποφάσεων προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις προθεσμίες έτσι όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και να προλαβαίνουμε έτσι να γνωμοδοτούμε. Πιστεύω απόλυτα ότι οι νέοι κανόνες μας προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο συλλογής αλλά και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με μακροεποπτικά μέτρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως πρώτο βήμα Έχουμε ήδη καθορίσει ένα χώρο στην ιστοσελίδα μας όπου θα δημοσιεύουμε όλα τα εθνικά μέτρα τα οποία φτάνουν στην προσοχή μας σε σχέση με την πρώτη σύσταση που κάναμε όσον αφορά το δανεισμό σε ξενονόμισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας τώρα για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε σειρά παρεμβάσεων, ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα, Jean-Paul Gauzès. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω προηγουμένω, όπως προβλεπόταν. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε, συνεργασία της Επιτροπής μας του Κοινοβουλίου με εσάς και εφόσον αυτή η συνεδρίαση έχει την απόχρωση τέλους θητείας, παρόλο που ελπίζουμε να τα ξαναπούμε, εσείς θα είστε σίγουρα εκεί, εμείς λιγότερο σίγουρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια μαθήματα έχετε πάρει από πλευράς της βούλησης του Κοινοβουλίου. Δηλαδή να γίνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας, επίσημος πρόεδρος της Επιτροπής, μετά από το χρόνο αυτό τη θητεία μπορεί να μα πει ήταν η ιδέα, ήταν καλή, έπρεπε να συνεχιστεί ή αν πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. I'm not sure I got the end of your questions. It said... Κατάλαβα τις ερωτήσεις. Τι μαθήματα μάθαμε από το Κοινοβούλιο. If Ίσως προ... ήθελα να μιλήσω γρήγορα για να κερδίσω χρόνο. Θα ήθελα να ξέρω το εξή. Αποφασίστηκε όταν δημιουργήθηκε η Επιτροπή ότι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι και πρόεδρο τη εν λόγω Επιτροπή τουλάχιστον κατά την αρχική φάση. Και πέρασε κάποιο χρόνο. Έχετε κάποια εμπειρία. Λοιπόν, εξ αυτού, ποια μαθήματα έχετε συναγάγει για την κατάσταση. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση ή να ακολουθήσουμε άλλες διαφορετικές πρακτικές. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ο κ. Αλκαντράουι έχει το λόγο. είσαστε σε περίεργη θέση, δεν σας βλέπω γιατί έχω από πίσω τον ήλιο παρόλο που έχει την κουρτίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Καντράη, για, τους, για την αγορά νομισμάτων, για την αγορά χρήματος. Έγιναν κάποιες συστάσεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρότεινε λοιπόν για την αγορά χρήματος έναν κανονισμό για να αντιμετωπιστεί οι ε, τραπεζικές διαδικασίες. Και έγιναν συστάσεις από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου τέλος 2012 μαζί με το Εθνικό Νομισματικό Ταμείο. Ζητήθηκε υποχρεωτική μετακίνηση προς, προς τα βίναυς. Σαν εισηγητής πρότεινε ένα συνδυασμό των προτάσεων αυτών αυτό που πρότεινε, δηλαδή ένα περιθώριο προστασίας, buffer, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια μετατόπιση προς τα VNAVs σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας κάποια μέλη αμφισβητούν την ανάγκη που υπάρχει και τον κατεπίγοντα χαρακτήρα αυτής της ανάγκης για λήψη συμπληρωματικών μέτρων όσον αφορά τα VNAVs. Ερώτηση. Επιβεβαιώνεται τη θέση της, του Ευρωπαϊκού ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Μάλλον Συστημικού Κινδύνου για τα Βίναυς και πώς μπορούν να αποφύγουμε τους κινδύνους των ΖΙΝΑΒΣ και κυρίως πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από τα ΖΙΝΑΒΣ προς τα ΒΙΝΑΒΣ. Πώς απαντάτε σε αυτούς με τους οποίους δεν συμφωνώ που φοβούνται ότι αυτό το buffer ή αυτή η αλλαγή από το ένα σύστημα στο άλλο θα είναι κάτι αντιπαραγωγικό. Ότι θα δημιουργήσει και άλλους κινδύνους διότι τα χρήματα που είναι στα ταμεία θα πάνε στις τράπεζες ή και ίσως και τα χρήματα αυτά να βγουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Συλλέγουμε τις ερωτήσεις λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Μπούλς. Σιλβί, θέλεις να πάρεις το λόγο ή όχι. Να πω ότι σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρουσία σας, λέει η κυρία Γκουλάρ. Και εγώ ρωτώ όπως ο κύριος Γκοζές για το ρόλο σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την άλλη ερώτηση για τα ΖΙΝΑΒΣ και τα ΒΙΝΑΒΣ και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ η Βίκη Φόρντ για το ECR έχει το λόγο. Είναι βαρετό ερώτημα αλλά σημαντικό διοικητικά. Ελπίζω να μην με κάνει γραμματέα του James Bond αυτή η ερώτηση. Κυρία Μόνη Πένη. Περάσαμε πολύ χρόνο προσπαθώντας να σπάσουμε το φαύλο κύκλο που οι φορολογούμενοι γλιτώνουν τις τράπεζες, διασώζουν τις τράπεζες. Λοιπόν, δημιουργήσαμε αυτό το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για, την, για το συστημικό κίνδυνο, φέραμε τους καταθέτες σε προτιμησιακή θέση, και εν μέρη επίσης βρήκαμε λύση μέσω του σημαντικού ρόλου που, παίζει, που παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την, τους κρατικούς ενισχύσεις. Όσον αφορά το ESRM δώσαμε πολλούς νέους ρόλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν του αρχικού ρόλου e SRM και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και αυτό είναι μια ανησυχία διότι το θέμα των κρατικών ενισχύσεων είναι σημαντικότατο όσον αφορά την προστασία του χρήματος των φορολογωμένων και την αποφυγή κινδύνων. Όταν δημιουργήσαμε αυτό το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, σαν Κοινοβούλιο υπήρξαμε σαφέστατοι. Θέλαμε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των ρόλων σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Θέλαμε ξεχωριστές γραμματείες, ξεχωριστό προσωπικό τι συμβουλή δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αποφυγή της συγκρούσεως συμφερόντων. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα η προστασία του χρήματος των φορολογωμένων και να μην υπάρχουν ηθικά δεντολογικά προβλήματα και να αποφύγουμε τις χρεοκοπίες των τραπεζών. Jean-Paul για τους Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός, κάτι που συστήνεται, λέει Μπεσέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχέση με αυτά που προαναφέρθηκαν. Ποια είναι η άποψή σας για τις σοβαρές αναταραχές των αγορών των αναδιωμένων χωρών τους τελευταίους μήνες, κάτι που απειλεί ε, με επανεμφάνιση. Αυτές οι αναταραχές δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, για τις οικονομίες του κόσμου και κυρίως για τις ευρωπαϊκές οικονομίες που βασίζονται πολύ στην ανάπτυξη των αναδειωμένων αυτών χωρών. Δεν δείχνουν αυτά ένα νέο, μια νέα οικονομική καταιγίδα με συνέπειες καταστροφικές ενδεχομένως. Ανησυχούμε λόγω ενδεχόμενης συστολής μειώσεως της ζωής των κεφαλαίων και των πιστώσεων στις αναδιόμενες χώρες. Αυτό θα είχε αρνητικότατες συνέπειες όσον αφορά την εσωτερική ζήτηση των χωρών, άρα και επί των οικονομικών δραστηριοτήτων των οικονομιών της Ενώσεως. Ανησυχούμε πολύ περισσότερο, διότι μία από τις θεμελιώδεις αιτίες αυτής της κρίσεως, δηλαδή η σταδιακή εγκατάλειψη της πολιτικής της ελαστικής των διαφόρων κεντρικών τραπεζών, η επιβράδυνση της πολιτικής ενεργού εξαγοράς ίσως να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, να το πούμε διαφορετικά, δεν θα έπρεπε να προετοιμαστούμε για να αποφύγουμε εκπλήξεις όπως εδώ και πέντε χρόνια. Η Επιτροπή του Συστημικού Κινδύνου ετοιμάζεται για όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Ευχαριστώ. Καλώς για την ΚΟΕ η Μαρίζα Ματέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, θα ήθελα θα ήθελα με την ευκαιρία της δεύτερης αυτής συζητήσεως να έρθω σε ένα θέμα που είναι, εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρο. Δηλαδή τον τραπεζικό κίνδυνο και τον κίνδυνο των κρατικών ομολόγων που εξακολουθούν και είναι πολύ παρόντα. Και σε σχέση και με την ερώτηση που έθεσα προηγουμένως για την έκδοση δανείων από τα κυριότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο η έλλειψη πρόσβασης σε πίστοση, αλλά και η έλλειψη ζητήσεως, που έχει σχέση όμως και με τις βαριές πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν στην καταβαράθρωση των μισθών. Και εγώ νομίζω ότι φέρεται μεγάλη ευθύνη εκεί. Όμως η σχέση μεταξύ ε, τραπεζικού κινδύνου κοινού των τραπεζών δηλαδή και του κρατικού δανεισμού. Οι τράπεζες και τα κρατικά ομόλογα παραμένουν συνδεδεμένα. Οι τράπεζες εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία έχουν τρέδρα έδρα και από την πολιτική επιτοκίων. Οι Πορτογάλοι σε σχέση με τους Γερμανούς πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερο επιτόκιο, 5,5% ενώ στη Γερμανία είναι 3,6%. Είναι λοιπόν περίπου 60% περισσότερα αυτά που πρέπει να πληρώσουν οι Πορτογάλοι επιχειρηματίε για να χρηματοδοτηθούν από τι τράπεζε. Όταν θα κάνετε τι δοκιμασίε αντοχή, η ιδέα είναι να προσπαθήσετε να μειώσετε και την σημασία του, του παράγοντα της έδρας, τον τοπικό παράγοντα δηλαδή. Όμως τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε μεγάλη δυσκολία να φτάσετε σε ολοκλήρωση του μηχανισμού εξυγίανσης τραπεζών, διότι όσα έχετε κάνει για να ξεπεραστεί ο παράγοντας του τόπου δεν λειτουργούν. Τα ίδια φαινόμενα βλέπουμε και αλλού. Τα, οι δοκιμές αντοχής δεν θα έχουν καμία επίπτωση τελικά στην πρόσβαση σε πίστη των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Μέγα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κύριε Πρόεδρε, και ο χρόνος που σας διαθέτω είναι όσο χρειαστείτε. Θα ακολουθήσω τη σειρά με την οποία τέθηκαν οι ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στον ρόλο του ESRB από τότε που άρχισε να λειτουργεί. Στρέφοντας τα βλέμματα προς τα πίσω, ο ESRB δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε ως παρουσία μέσα στον συνεχιζόμενο λόγο για τον δημοσιονομικό κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε τη δουλειά του ESRB σε δύσκολο περιβάλλον, γιατί θα θυμάστε ότι η κρίση μόλις είχε ξεσπάσει και συνέχισε τη δουλειά του μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον όπου αναφύονταν νέοι οργανισμοί, νέοι θεσμοί και νέες δραστηριότητες. Όταν έγινε ο ESRB δεν υπήρχε ούτε SSM, ούτε SRM, ούτε προοπτική να γεννηθούν. Και πολλά από τα βήματα που λήφθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια επίσης δεν είχαν δεν προβλέπονται να γίνουν. αντιμετωπίσαμε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που προσαρμόστηκε αρκετά καλά διατηρώντας το ρόλο του, υπακούντας την εντολή του ε, για το περιβάλλον αυτό και με τα χαράς ήμουνα πρόεδρος του SRB και θα κάνω ό,τι μπορώ για να κατευθύνω αυτό το όργανο μέσω των αναγκαίων αλλαγών του των λεχθέντων η εντολή μου είναι στα χέρια σας κατά κάποια έννοια, στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τώρα επιτρέψτε μου να πω εν γέννη ότι αν δω ε, ποια είναι η βάση, που κινείται η βασική γραμμή στην οποία κινείται το SRB και ποια είναι τα αποτελέσματα, είναι θετικές εντυπώσεις. Πάμε στο δεύτερο σημείο για, για την αγορά χρήματος και τα σχετικά ταμεία. Θα σας πω ότι θα θυμόσαστε ποια ήταν η θέση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Δηλαδή, θέλαμε να σχεδιάσουμε την σύγκληση των ταμείων σύναφ σε ταμεία βίναυ υποθέτοντας, ο, υποθέτοντας συμπεραίνοντας ότι το σύναυς εμπεριείχε συστημικό κίνδυνο. Αυτό ηρίσταν παρόδο ήταν και η θέση του ΦΕΔ των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό δεν σημαίνει ότι είπα θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, διότι η SEC φαίνεται ότι έχει διαφορετικέ απόψει. Άρα υπάρχει α, ποικιλία απόψεων. Η συζήτηση του SRB έλαβε χώρα πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει την πρότασή τη για ένα 3% ε, περιθώριο κεφαλαίων για τα σύναυς για κάποια χρονική περίοδο και μετά αυτή την περίοδο θα μετατραπούν σε βίναυς δεν είχαμε συζήτηση στο ESRB για το πώς θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά πρέπει να πω ότι καταρχάς από μια πρώτη άποψη θα ήταν μια δεύτερη θέση αν θέλετε, δεύτερη λύση σαν βήμα προόδου. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου του Συμβουλίου διότι δεν διεξήχθη η συζήτηση ακόμα. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή ότι θα είναι ένα δεύτερο βήμα, δεύτερο σε σημασία, αν θέλετε δεύτερο καλύτερο βήμα πρόοδου. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την ίδια αξιολόγηση όπως το, το ε, Επιτροπή Στημικού Κινδύνου όσον αφορά τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα σύναυς. Το 3% το όριο του 3% είναι τελικά ίσως κάτι που δεν έχει νόημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δαπανηρό και το μέσο θεωρεί κάτι πολύ δαπανηρό. Το τρίτο ερώτημα όσον αφορά τις αναταραχές της διαταράξεις αυτές. Αυτές τις αναταράξεις στις χρηματοψηφιστικές αγορές Αναφέρεστε στα σημερινά γεγονότα ή γενικότερα σε αυτά που συνέβησαν τους τελευταίους ε, μήνες. Εάν αναφερόμαστε στα σημερινά γεγονότα, είπα πριν ότι αν δούμε ποσοτικά τι σημαίνουν αυτά, αν δούμε τι, πώς επηρεάζουν τον εμπορικό τομέα και πώς επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, παρόλο που δεν βλέπουμε σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι είναι δυσχερέστατο να προβλέψει κανείς τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνέπειες τέτοιων μεγάλων γεωπολιτικών κινδύνων. Όμως, αν αναφέρεστε στις αναταράξεις των τελευταίων μηνών, θα έλεγα ότι η Ευρωζώνη σε μεγάλο ποσοστό τα κατάφερε πέρασε από τις αναταράξεις αυτές με θετικό τρόπο. Η αντίδραση στα προβλήματα που συνέβησαν στη ΣΥΠΑ ήταν θετικά. Πολλά είχαν κοστολογηθεί ήδη στην αγορά. Όσον αφορά την Ευρωζώνη, ο αντίκτυπος δεν είναι αρνητικός. Μάλιστα θα έλεγα ότι οι αποδόσεις των μετοχών στις χώρες δοκιμής αντοχής ήταν κάτι χαμηλό μετά την παρέμβαση που έγινε στις Πολιτείε. Υπάρχουν όμως συνέπειες όσον αφορά τις αναδυόμενες οικονομίες και εκεί η απάντηση είναι θα έλεγα αρκετά περίπλοκη. Έχουμε τρεις, τριών ειδών, τρεις κατηγορίες φορέων. Το σημαντικότερο φορέα που είναι οι κυβερνήσεις των ίδιων των αναδυομένων αγορών βλέποντας τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα όσον αφορά τις οικονομίες των αναδιωγμένων αυτών χωρών, βλέπουμε ότι περισσότερο πλήγουν τις πλέον ευάλωτες οικονομίες. Οι οικονομίες που είχαν πολύ μεγάλο έλλειμμα στον προπολογισμό και στον τρέχοντα ισολογισμό μεγάλα ελλείμματα, υψηλά επίπεδα εν γέννη, ε, χρέου και πολύ χαμηλά αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενετόπισε πέντε ευάλωτες ε, χώρες. Άλλες αναδιόμενες χώρες τα κατάφεραν, αντιμετώπισαν ε, αυτά τα προβλήματα με καλύτερο τρόπο Άρα η πρώτη ομάδα φορέων είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που θα πρέπει να κάνουν πιο ανθεκτικές τις οικονομίες τους μέχρι μέσω σωστών οικονομικών πολιτικών. Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς, άλλη ομάδα φορέων που είναι οι κεντρικές τράπεζες ή οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές δικαιοδοσίες. Μεγάλοι φορείς. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται αυστηρό συντονισμό. Μάλιστα, αυστηρό συντονισμό μεταξύ μα είναι δύσκολο, διότι κινόμαστε εντό εθνικών ορίων και εντολών. Όμω πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι οι δράσει μα συνεπάγονται συνέπειε προ αναδυόμενε αγορέ και θα πρέπει αυτό να το παραδεχτούμε και το λάβουμε υπόψη μα στη διαμόρφωση νομισματικών πολιτικών μα. Υπάρχει και τρίτο τομέα φορέων που μπορεί να κάνει τα περισσότερα. Σε όλα αυτά οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπορεί να βελτιώσει την αντοχή των αναδειωμένων οικονομιών ποικιλοτρόπος. Ρίσταν παρόδο ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτές οι χώρες είχαν στη διάθεσή τους το FCL όπως αποκαλείται και δεν το χρησιμοποίησαν λόγω του φόβου του στίγματος ότι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πιστώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει το Δούνο του όσον αφορά τον περιορισμό των συνεπειών που έχουν οι νομισματικές αποφάσεις που λαμβάνονται εντός των διαφόρων ε, αρμοδιοτήτων. Μετά. Τελευταία ερώτηση. Η σχέση μεταξύ τραπεζικού κινδύνου, αν με Κάτι άλλο, ναι, ναι. Αν κατανοώ καλά την ερώτησή σας, έχει να κάνει με την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως διαχειρίστριας της κρατικής, των κρατικών επιδοτήσεων. Η ερώτησή μου είναι πώς διαχωρίζετε τους δύο ρόλους. Πώς λέτε την σύγκρουση συμφερόντων αφενός μεταξύ της κρατικής επιχορήγησης και αφετέρου της εξυγίανσης των τραπεζών. Τι έχει λειτουργήσει και τι όχι κατά τη γνώμη σας εκεί. Κοιτάξτε, πρόκειται για μέρος της, της του SRM που θα πρέπει να έχει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να αποφασίζει με τρόπο βέβαια συμβατό με τους κανόνες για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Να είναι όμως ανεξάρτητο Συμβούλιο, να μπορεί να λαμβάνει ταχαίως αποφάσεις και ανεξάρτητα. Ας μην λησμονούμε ότι και στο εθνικό επίπεδο, εάν εξετάσουμε τις αρχές εξυγένσης των τραπεζών στο εθνικό επίπεδο, ή αν θα έχουμε μία ενιαία τέτοια αρχή. Οι προβληματισμοί τους θα πρέπει να είναι συμβατοί με τους κανόνες των κρατικών επιχορηγήσεων για να αποφευθεί ο φορολογούμενος να επιδοτεί το τραπεζικό σύστημα. Μα θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία Φόρντ, τον τελευταίο λόγο και για την εξυγίανση και για την resolution και για τις κρατικές επιχορηγήσεις ώστε η ανεξαρτησία εδώ για την απόφαση για τις κρατικές επιχορηγήσεις ενδεχομένω να τίθεται σε κίνδυνο. Γι' αυτό και ρωτώ η εμπειρία σας ποια, είναι. Κοιτάξτε, στην περίπτωσή μας η νομισματική πολιτική διαχωρίζεται ξεκάθαρα από την εποπτεία με ένα πλήθος κανόνων και τώρα ε, φτιάχνουμε μάλιστα και ένα εσωτερικό εγχειρίδιο διαδικασιών. Επειδή εγώ ήμουν στην ίδια κεντρική τράπεζα και διοικητής και επικεφαλής της εποπτείας, οι συγκρούσεις αυτές συμφερόντων είναι δυνατόν να, τις διαχειριστούν με το σωστό διαχωρισμό και του ίδιου είδους διαχωρισμός μπορεί να επιβληθεί και στο νέο SRM ανάμεσα στους δύο ρόλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως είναι σωστό αυτό που λέτε και πρέπει να το παρακολουθούμε για να διασφαλίσουμε ότι όντως θα συμβεί αυτό, ο διαχωρισμός δηλαδή. Η τελική ερώτηση είχε σχέση με την σχέση με τον κίνδυνο των τραπεζών και των κρατικών ομολόγων. Πρώτα, να το εξετάσουμε αυτό με μια προοπτική. Ο σύνδεσμος αυτός που αποκορυφώθηκε το 2010. Αγνοήθηκε πλήρως, είχε αγνοηθεί μάλλον πλήρως μέχρι να ξεσπάσει η οικονομική κρίση και ήρθε σε, πλήρως, σε πλήρες φως με το PSI, το κούρεμα δηλαδή. Τώρα έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τις τράπεζες. Έχει λοιπόν υποχωρήσει. Όχι εντελώ όμως. Ξεκολουθεί και υπάρχει κατακαιρματισμό από την πλευρά του δανεισμού, όπως είπατε και πριν, αλλά και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, αν εξετάσετε πώς επενδύουν οι ασφαλιστικές εταιρείε τα αποθεματικά τους ασφαλιών ζωής, θα δείτε ότι είναι οι επενδύσεις αυτές κατακαιρματισμένες δηλαδή επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία της ίδιας χώρας όπου βρίσκονται οι ασφαλισμένοι τους. Και μπορεί να εξετάσει κανείς και πολλές άλλες πλευρές του κατακαιρματισμού αυτού και αν το εξετάσει κανείς πρέπει να ε, δει ότι κάνει, πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες ακόμα για να ξεπεραστεί ο κατακαιρματισμός αυτός. Η δημιουργία του SSM σημαίνει μια ακόμα μείωση του συνδέσμου αυτού αποδυναμώνει τον σύνδεσμο αυτό ακόμη περισσότερο διότι η αξιολόγηση των τραπεζών στις διάφορες στα διάφορα μέρη της Ευρώπης θα γίνει από ένα κοινό επόπτη. Θα υπερβαίνει δηλαδή τον εθνικό επόπτη και τις υποψίες που ενδεχομένω θα προκαλέσει μια καθαρά εθνική εποπτεία που ίσως να επηρεαστεί από επενδυμένα συμφέροντα που έχουν την έδρα του στη χώρα αυτή. Τώρα βέβαια τούτου λεχθέντος Πλήρη στράψη του συνδέσμου μεταξύ των δύο μπορεί να επιτευχθεί μοναχά με τη, με δημιουργία του SRM, του ενιαίου μηχανισμού εξηγένσης των τραπεζιών. Άρα προχωρούμε κατά βήματα. Είναι ήδη βελτιωμένη η κατάσταση απέναντι στην κατάσταση που ήταν τρία χρόνια πριν. Ο μηχανισμός SRM, μάλλον ο SSM ήδη αποτελεί ο νέος μηχανισμός υποπτία είναι ένα βήμα εμπρός και μάλλον το τελικό ρήγμα θα προκύψει από την εφαρμογή του SRM. Μάλιστα, εδώ ολοκληρώνουμε την συνεδρία αυτή, λέει η πρόεδρος Bowles και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, μιας και εμείς υποπτεύουμε εσά. Βεβαίως και θα ξαναειδωθούμε τις επόμενες εβδομάδες, όμως σας ευχαριστώ και πάλι όλος ιδιαίτερος. Okay. And I can just tell you our next meeting. Τώρα, η επόμενη συνεδρία μας θα είναι στις 10 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. We now need those who are coming to another meeting need to come quickly.